Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε εδώ συνάδελφοι και συνάδελφοι. Συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνάδελφοι από, το Εθνικό, από τα Εθνικά Κοινοβούλια και εκτιμώ όλου ιδιαίτερω την παρουσία σα εδώ. Αντιλαμβάνομαι βέβαια πόσο μεγάλη σημασία έχει και η κοινοβουλευτική συνέλευση. Εγώ είμαι στην ε, αντιπροσωπεία αυτή από τότε που είμαι ευρωβουλευτής από την Ελλάδα, εδώ, 7 χρόνια δηλαδή και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της επιρροής του ΝΑΤΟ έχει να κάνει πολύ και με τη συμμετοχή της Ευρώπης και με τις δικές σας προσπάθειες που όλοι μαζί προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των χωρών μελών, μεταξύ τους και με άλλους. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μπορούμε να λύσουμε πράγματα που αλλιώ θα ήταν ίσως πολύ πιο δύσκολο ή αδύνατο να λυθούν. Εκ μέρου λοιπόν τώρα της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπεία Αντιπροσωπείας ε, στο ΝΑΤΟ, ε, Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να καλωσορίσω εδώ θερμά τον Αντιπρόεδρο Πάσκου, ο οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας. Ε, Επίσης έχει ντοκτορά σε πολιτικές επιστήμες και να σας διαβάσω τώρα το βιογραφικό του, δεν θα είχε χρόνο να πάρει το λόγο εκείνο. Είναι όμως πραγματικά τιμή που τον έχουμε αντιπρόεδρο εδώ υπεύθυνο για τις δραστηριότητές μας. Καλωσορίζω επίσης θερμά και όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση υψηλού επίπεδου. 20 μέλη από 14 χώρες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και επίση καλωσορίζω θερμά εδώ και τον πρόεδρό τη, τον Παόλο Άλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα συμπροεδεύσουμε σήμερα. Η δικιά του πρόταση ήταν να λάβει χώρα η εκδήλωση αυτή σήμερα. Είναι από την Ιταλία και ίσως και γι' αυτό είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος όσον αφορά τις χώρες μέλη που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Ε, στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, είναι γνωστό, μπορεί να μην είναι ακριβώς άμυνα, αλλά είναι πολλές και διαφορετικές που έχουν να κάνουν όμως με την ασφάλεια. Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λοιπόν με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικές και τονίζω πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι κοινοβουλευτικοί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προστατεύουν τους πολίτες, αλλά προσφέρουν και διατλαντική αλληλεγγύη. Δεν έχουμε ακόμα όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Θα ενισχυθεί όμως αυτή η σχέση όλο και περισσότερο. Επίσης, μπορέσαμε να συμμετέχουμε ως Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ τον Παόλο Άλλη και τους συναδέρφους του για την εξωτερική οργάνωση της διάσκεψης ε, της Ερηνής είναι καλό να μπορούμε να ε, συμμετέχουμε και να προβάλλουμε τη συνεργασία αυτή όλο και περισσότερο. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι όλο και πιο περίπλοκες. Υπάρχουν νέες ε, απειλές που μπορεί να είναι από κρατικούς παράγοντες, από μη κρατικούς παράγοντες, υβριδικές σημεί, από νότια, από ανατολικά, που θέτουν ε, θέματα καινούρια. Νέες απειλές και πιο περίπλοκες απειλές απαιτούν όλο και περισσότερο συνεργασία και κοινέ λύσεις και κοινή δράση. Πρέπει συνεπώς να διαβρύνουμε ακόμα περισσότερο την στρατηγική αυτή εταιρική σχέση μεταξύ μας, να έχουμε περισσότερες ικανότητες περαιτέρω και να αποφεύγονται επικαλύψεις δράσεων και δομών. Όσο γίνεται βέβαια αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δαπανίσουμε πιο αποτελεσματικά τα κονδύλια που διαθέτουμε και οι κοινοβουλευτικοί το θεωρούν αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο του δεσμού τη κοινοβουλευτική διάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και πιστεύω ότι θα συνεισφέρει και στην επόμενη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο που θα συναντηθούμε πάλι εκεί και αναμένουμε βέβαια να υπογραφεί και νέα κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ε, θα έλεγα ότι οι ε, εταίροι μας πρέπει να είναι ασφαλείς, πρέπει να φροντίσουμε για την προστασία τους και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Και το λέω αυτό προερχόμενοι από μια χώρα που αντιμετωπίζει και οικονομική κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν δώσω το λόγο στον Παύλο πάντως για τις αγωγικές του παρατηρήσεις, να ξέρετε ότι έχουμε διερμηνία στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πολωνικά, ολλανδικά, ελληνικά, σουηδικά, τσεχικά, κροατικά και τη γλώσσα του Μαυροβουνίου. Ε, πρόκειται για δημόσια συνάντηση, η οποία θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Υπάρχει καφές, τσάι, ό,τι θέλετε, για μερικές ώρες ακόμα εδώ στο τραπεζάκι. Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Και τώρα που έχετε νέα κυβέρνηση στην Ιταλία, περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα τους επόμενους μήνες, τι θα σημαίνει αυτό για την Ευρώπη επίσης. Πάντως, συγχαρητήρια για την τόσο πετυχημένη εκδήλωση που οργανώσατε. Ευχαριστώ, Εύα, για την εισαγωγή και για το γεγονό ότι μας φιλοξενείτε εδώ σήμερα. Όπως ε, γνωρίζετε και όπω είπατε, ένα από τα θέματα τα οποία αποτέλεσε προτεραιότητα της Προεδρίας μου ήταν να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών οργανισμών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, πρωτίστως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεργαζόμαστε από αυτού και με την πλήρη στήριξη του Προέδρου Ταγιάννη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συνάντηση και αυτός είναι ένας τρόπος να καταδείξουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ κοινοβουλευτικών ε, οργανισμών, γιατί πιστεύουμε ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο συμπληρώνει την κυβερνητική διπλωματία και το βλέπουμε σε κάθε επίπεδο των δραστηριοτήτων μας. Και με καθησυχάζει το γεγονός ότι βλέπουμε εδώ μια ομάδα νομοθετών και αξιωματούχων από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες εταίρους. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ε, αναπλοηρότρια Γενική Γραμματεία, την κυρία Κοτερμίλη, μόλι έρθει και τον κύριο Σεράνο από την ε, Κοινή Υπηρεσία Ασφάλεια και Άμυνα όταν θα έρθει. Επίση, να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του ε, δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων ε, που πάντα ήταν πολύ σημαντική ε, σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και ΝΑΤΟ και τα προγράμματα προσέγγισης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα η όθηση έρχεται από νέε και σύνθετες προκλήσεις για την ασφάλεια, οι οποίες αναδύθηκαν και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο την τελευταία τετραετία. Τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, αποστεθεροποίηση, μεταναστευτικά κύματα, διάφορες απειλές όπως αναφέρατε προηγουμένως, κυβερνοεπιθέσεις, ε, πολιτικές παρεμβάσεις, ε, ε, παράνομη ε, προσάρτηση εδαφών, ε, κατάληψη εδαφών από την Ρωσική Ομοσπονδία που συνεχίζουν να ανησυχούν τον ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή αντίληψη της ευρωπαϊκής σταθερότητας το νέο περιβάλλον ασφαλείας ε, και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει προσαρμογή. Και οι δύο μιλούν για νέα καθήκοντα και αποστολές, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και την κατάλληλη ισχύ να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις σε μη παραδοσιακές επιθέσεις με νέα εργαλεία και νέα μέσα. Και πρέπει να προσέξουμε και τι πόρους χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των νέων ευθυνών. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας ως Ευρωβουλευτές ε, να κατανοήσουμε ότι δεν ε, είναι μόνο το πλαίσιο, αλλά και η αξία των προτινόμενων λύσεων που έχει σημασία. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να υποστηρίξουμε την κατάλληλη άγουσα και να υπάρχει κατάλληλη δημοκρατική υποστήριξη για να τα υποστηρίξουμε σε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς ε, σε όλη την Ευρώπη. οι σημερινές ε, προκλήσεις ασφαλείας, ε, κυρίως ε, εδώ στην Ευρώπη, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει αποφασιστική συμβολή από τους συμμάχους και τους εταίρους και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας οργανισμός που μπορεί να τα χειριστεί όλα μόνος του. Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυσική εταίροι ασφαλείας. Υπάρχουν 22 κοινά μέλη και έχουμε πολλές κοινέ αξίες οι οποίες καθορίζουν και τις αρχές των κρατών μελών και φυσικά και πολλά κοινά στρατηγικά συμφέροντα. Όπως γνωρίζουμε βεβαίως, έχει υπάρξει πολύ ψηλός βαθμός ε, επιφυλάξεων στο παρελθόν για το πώς η συνεργασία θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αναφερθήκατε σε επικαλύψεις, σε όλες αυτές τις ανησυχίες για τα θέματα αυτά. Αλλά Νομίζω ότι η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που επιβεβαιώνει το ρόλο του ΝΑΤΟ ως ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας ε, και η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά από την ε, παραδοχή ότι υπάρχει ένα σύνολο δυνάμεων είναι πολύ σημαντική. Η Σύνοδος της Βαρσοβίας το 2016 ξεκίνησε μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και οι πρωτοβουλίες που θα συζητηθούν σήμερα εδώ σαφώς θα αποδείξουν ότι όντως ξεκίνησε μια νέα εποχή. Υπάρχουν βασικοί τομείς, επτά τον αριθμό, που ε, είναι πολύ φιλόδοξοι για τον καθορισμό της στρατηγικής, αλλά αυτές οι πρωτοβουλίες χρειάζονται όλη την υποστήριξη που μπορούμε να έχουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό είστε όλοι εδώ σήμερα η ε, κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η εταιρική του σχέση είναι καλός τρόπος για να ε, το επιτύχουμε αυτό και ενισχύει τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Σύνοδο της Βαρσαβίας και μετά. Σε λίγους μήνες θα συναντηθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από τους βασικούς τομείς της Συνόδου είναι η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας πριν από μερικές ημέρες ε, στη Σύνοδο ε, της Βαρσοβίας, στην Νεαρινή Σύνοδο. Η παρουσία μας εδώ σήμερα θα αποστείλει ε, σίγουρα ένα στεναρό μήνυμα υποστήριξης, ε, κάτι το οποίο είναι σαφές και στη δήλωση και επιβεβαιώνει την ενότητα και την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο των Βρυξελών, η οποία εγκρίθηκε πριν από μερικές ημέρες στη Βαρσοβία. Ε, πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική για το συντονισμό των δυνάμεων των δύο οργανισμών, διότι μέσω της προσαρμογή θα επιβιώσουμε, αλλά ταυτόχρονα θα βρούμε και τα μέσα για να ξεπεράσουμε τις νέες προκλήσεις ε, που ε, μας... Ε, αφυπνίζουν και να μην υπάρχουν διαιρέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε και τα θέματα ασφαλείας, ε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προκλήσεις και, από, και εκ των έσω. Και ελπίζουμε να έχουμε και πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ε, σύντομα ε, ελπίζω για κοινή ασφάλεια και άμυνα στην Ευρώπη, ώστε να έχουμε και ισχυρότερη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε ο Άλσεντε Ντεγάσπαρη πριν από 70 χρόνια. Εάν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν κοινά σύνορα και τα οποία πρέπει να υπερασπιστούμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης και ότι υπάρχει εντός των σύνορων είναι και μια κοινότητα εθνών. Δεν είναι ε, ανεξάρτητες και ξεχωριστές χώρες. Η ισχυρότερη πολιτική ένωση λοιπόν απαιτείται αυτή τη στιγμή ενώπιον μιας πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, η οποία αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε και πολιτική αστάθεια, αντιφάσεις, αυξανόμενο λαϊκισμό. Δείτε ε, πως ε, κάποια θέματα όπως η μετανάστευση και η διαφθορά ε, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης των λαϊκιστών και έχουμε απτές αποδείξεις της αστάθειας σε αρκετές χώρες, χώρες οι οποίες παραδοσιακά ήταν πολύ σταθερές, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, στην Ιταλία, ο Σαλβίνη κλπ. Και τώρα τι θα γίνει με το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν θα πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να αφήσουμε τις παρούσες διαφωνίες μεταξύ μας, οι οποίες υπάρχουν, να αποδυναμώσουν την εταιρική μας σχέση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ισχύς εν του ενώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την ε, προσοχή σας και την πρόσκληση και εύχομαι μια καρποφόρα ε, ημέρα για όλους. Thank you ευχαριστούμε πάρα για τα εξαιρετικά σας σχόλια. Νομίζω πως ε, οι χώρες μας, η Ελλάδα και η Ιταλία, είναι ε, χώρες όπου παρατηρείται ε, ένας φόβος για το άγνωστο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες εν ώψη εκλογών. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω μία ακόμα φορά τον κύριο Πάσκο, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής σχέσεων με τα πολυμερή όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΑΤΟ. Δραστηριοποιείται όμως σε πολλούς περισσότερους τομείς και πρόσφατα κατάρτισε μια έκθεση αρκετά περιεκτική για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Πριν, λίγες εβδομάδες πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ασχοληθήκαμε και με την συνεργασία ανάμεσα με τους δύο οργανισμούς. Σας δίνω λοιπόν το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. Ευθύς Σας ευχαριστώ πολύ. αισθάνομαι πως ε, βρίσκομαι σε μια συναυλία και πως είμαστε η μπάντα που θα προετοιμάσει το κοινό για το κύριο σχήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι προέρχεστε και εσείς ήδη από τις από μεσογειακές χώρες, από την Ιταλία, από την Ελλάδα και με κάνετε να θυμάμαι μια περίπτωση Τη ρωσική αντιπροσωπείας που μόλις είχε φτάσει στο Βουκουρέστι μύρισε τον αέρα και αναφώνησε «Είμαστε στη Μεσόγειο». Και εμείς λοιπόν, και η χώρα μα είναι μεσογειακή χώρα. Και πιστεύω πως είναι πάρα πολύ θετικό ε, το γεγονός ότι δεν συναντιόμαστε μόνο σε αυτά τα ετήσια συνέδρια, αλλά και πολύ συχνότερα. Γι' αυτό λοιπόν, εκ μέρου του Προέδρου Αντώνιο Ταγιάννη, θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωση ε, ΝΑΤΟ εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μένα, όπως και για εσάς, είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή, ε, διότι η παρουσία και της ε, ρουμανικής αντιπροσωπείας είναι εδώ και είμαι αρμόδιος για αυτά τα θέματα από το 2000. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε για μένα, το έργο μας ε, και η ομαλή λειτουργία της συμμαχίας. Πρωτού συνεχίσουμε όμως, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στο θέμα τη σημερινή συνεδρίαση, την αντιμετώπιση νέων απειλών και τη νέα εποχή της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ένα μέρος αυτής της ε, αντιμετώπισης είναι η επανενεργοποίηση των λεγόμενων παλαιών απειλών τη στρατιωτική επιθετικότητας γειτονικών χωρών που, με την οποία ήρθαμε αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις, όμως να μην ξεχνάμε και τις παλιές. Υπάρχει, αν θέλετε, μία συνολική αντιμετώπιση. Πρέπει να το δούμε συνολικά. Οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί αρκετά και είναι λιγότερο προβλέψιμες και πιο επικίνδυνες. Υπάρχουν υβριδικές απειλές ε, που δημιουργούνται και από κρατικούς και από μη κρατικούς ε, φορείς και αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο και την ε, δυτική δημοκρατία. Μετά την μετά τον Σεπτέμβριο του 2013 όπου συζητήθηκε η σημασία της άμυνας Στόχος ήταν η προετοιμασία μιας νέας παγκόσμιας στρατηγικής για το 2016, η οποία και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από την ενίσχυση της διακυβερνητικής συνεργασίας, ε, στα πλαίσια του ΠΕΣΚΟ για παράδειγμα, όπως προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Ερευνών για την αμυντική βιομηχανία. Τώρα δημιουργείται μια, ένα νέο δεδομένο, δημιουργείται κοινή πρόσβαση σε κονδύλια για την άμυνα και δημιουργία κοινών προγραμμάτων άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πάντα ήταν πρωτοπόρος σε αυτές τις προσπάθειες και χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε πως οι προσπάθειές μας έχουν πλέον αντίκτυπο για παράδειγμα, ζητούσαμε νέα βιβλία για την άμυνα, ζητούσαμε νέες ε, επιτροπές, δημιουργία μιας γενικής διεύθυνσης άμυνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όπως αναφέραμε στην έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας το 2017. Όμως ε, δεν σταματάμε εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ήταν υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και καλωσορίζουμε την κοινή δήλωση των δύο οργανισμών ε, παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας στρατιωτικός οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι. Λειτουργούμε συμπληρωματικά και κοινό μα στόχο είναι η ειρήνη και η ασφάλεια. Η έκθεση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, την οποία παρουσίασε η πρόεδρο, όπως σας είπα, αναφέρει πως προσβλέπουμε στην νέα δήλωση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, η οποία θα εγκριθεί στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Η ενίσχυση και βελτίωση των υφιστάμενων προσπαθειών στην στρατιωτική συνεργασία, αναμυντική συνεργασία και ε, σε θέματα αμυντικής ε, βιομηχανίας και τεχνολογίας είναι πολύ σημαντική, καθώς και ε, η στήριξη χωρών ε, συμμάχων του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω μία ελπίδα και μία επιθυμία ότι θα καταφέρουμε στο μέλλον να συνεχίσουμε την ε, καλή δουλειά διατλαντικά παρά τα προβλήματάκια που μπορεί να έχουμε σε άλλους τομείς. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε τη σοφία που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε κάτι το οποίο μας προστατεύει όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να έχουμε ειρήνη είναι να διατηρήσουμε όσο έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τις πολύ καλές σας παρατηρήσεις, Αντιπρόεδρε, αλλά και για το έργο σας ε, γενικά που βοηθάτε να ενισχυθεί αυτή η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Είναι δύσκολο βέβαια να δουλεύει κανείς συγχρόνω σε πολλές υποθέσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μέλη και αντιπροέδρους που δραστηριοποιούνται πολύ. Δεν είναι αυτό κάτι που έχει γίνει πραγματικότητα πάντα, αλλά τέλος πάντων, γι' αυτό το εκτιμάμε όλου ιδιαίτερω. Τώρα, θα περάσουμε στο πρώτο θέμα που προβλέπει η ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας δεν είναι ακόμα εδώ. Θα έρθει όμως, έτσι. Οπότε θα δώσω σε εσά τότε πρώτα το λόγο. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω εδώ μία εξέχουσα μιλήτρια από τον μάλλον το μιλητή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης, τον κύριο Πέδρο Σεράνο, που είναι ο αναπληρωτής στην ε, Γενικός Γραμματέα ε, στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, ε, αντιδράσεις σε κρίσει κλπ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έτσι. Εξαιρετικός διπλωμάτης που προωθεί την εταιρική σχέση και τη συνεργασία και τους δεσμούς ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουλεύετε πολύ λοιπόν στο θέμα αυτό αντιμετώπιση των κρίσεων. Θα έλεγα τελευταία είμαστε μονίμως σε κρίση, έτσι δεν είναι. Ωραία, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βλέπω εδώ ότι ήρθε και η συνάδελφος, η Ρόζο Κιώτε Μουλέρ. Αλλά θα την αφήσουμε να προσγειωθεί θα κάνω εγώ την παρουσίασή μου και μετά εκείνη. Τώρα παίρνω το λόγο, για να μιλήσω ε, μετά. Πάντως και όσοι πήραν το λόγο πριν από μένα είναι ιδιαίτερα εξέχοντες και μίλησαν για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Με κάθε σεβασμό λοιπόν παίρνω το λόγο μετά τα όσα μας είπατε κύριε Πάσκου για την έκθεσή σας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει δίχως άλλο πάρα πολύ να αντιληφθούμε ακριβώς την μεγάλη σημασία που έχει αυτή η σχέση και να βρούμε την κατεύθυνσή μας για το μέλλον. Τώρα, όπως προβλέπετε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για νέες απειλές εδώ και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νέες απειλές που έφεραν πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ από ό,τι κατά το παρελθόν. Και αυτό έγινε και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συγχρόνως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζουμε τις δικές μας δομές ε, άμυνας. Δηλαδή θέλουμε ε, πιο ισχυρές ικανότητες άμυνας και αποτροπής, θέλουμε να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα από το παρελθόν ότι αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στην προσπάθειά μας πρέπει να συνεργαζόμαστε. Η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ είναι από τις πιο σημαντικές βέβαια όπως διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια και ευχαριστώ πολύ και την Ροζ Γκέντε Μούλερ και τους υπόλοιπους συναδέρφους για την τόσο καλή συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας. Δεν πρόκειται μόνο για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά είναι πραγματικά πολύ ευχάριστη συνεργασία με τους συναδέρφους αυτούς. Αν λοιπόν τώρα υπάρχει μια φράση που θα μπορούσε να συνοψίσει τα πάντα, είναι ότι μια πιο ισχυρή Ευρώπη είναι καλή για το ΝΑΤΟ και ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθώντα να πετύχουμε του στόχου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργαζόμενοι με το ΝΑΤΟ, ενισχύουμε και το ΝΑΤΟ. Είναι κάτι το οποίο έχει πει και επαναλάβει πολλέ φορέ και ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και η κυρία Μογκερίνη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ακριβώ είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε κι εμεί. Τώρα ένα στοιχείο κλειδί για τη συνεργασία μας είναι η κοινή δήλωση. Αναφερθήκατε ήδη σε αυτήν. Κοινή δήλωση της Βαρσοβίας του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟΥ και Προέδρου του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη συνεργασία με 74 δράσεις που πρέπει να υλοποιήσουμε. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τις 74 δράσεις. Η συνεργασία μας ξεπερνά τις 74 δράσεις. Τώρα έχουμε μια ε, διαδικασία συνεργασίας μεταξύ μας και του προσωπικού μας και όλες αυτές οι δράσεις δεν πρόκειται να εξαντλήσουν το θέμα, απλώς θα μας βοηθήσουν στη συνεργασία μας για να πετύχουμε κοινού στόχους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και οι Ρώσοι και άλλοι συνάδελφοι πολλές φορές μιλάνε για μια αλυσίδα νοτροπίας που ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για μια νοοτροπία καθημερινής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δεσμευτεί ε, μόνο, αν δεν δεσμευτεί μάλλον για τις δικές της ικανότητες, δεν βοηθάει τον ΝΑΤΟ. Άρα ούτε την ασφάλεια των πολιτών μας. Ένα λοιπόν από τα στοιχεία που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να ενισχύσουμε τις ικανότητες των χωρών μελών. Είναι στόχος κλειδί και για το ΝΑΤΟ. Το 2% στόχος που είναι οι αμυντικές δαπάνες βάσει του ΕΠ. Και στην Ουαλία το είπαμε αυτό. Και από τη δικιά μας την πλευρά η προσπάθειά μας βέβαια διαμορφώνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, αλλά βασικά είναι η ΠΕΣΚΟ, η συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα, που περιλαμβάνει δεσμεύσεις και ποιες είναι αυτές, να δαπανώμε περισσότερα για την άμενα, από κοινού, ανάπτυξη ικανοτήτων, είναι οι υποσχέσεις, δηλαδή δεσμεύσεις κλειδί που έχουμε πάρει εμείς βάσει της μόνιμης αυτής συνεργασία μας. Και έπειτα υπάρχουν και ειδικά προγράμματα τα οποία προσπαθούν να οδηγήσουν την πολιτική αυτή βούληση στην πράξη και στηρίζονται όλα αυτά από παράλληλες προσπάθειες που κάνουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της έρευνας με συγκεκριμένα προγράμματα και ελπίζουμε ότι θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια το χρόνο βάσει των νέων πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτή λοιπόν είναι η οικονομική ικανότητα και στηρίζεται και από ένα μηχανισμό αναθεώρησης που θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε κατά πόσο τελικά επιτυχάνουμε πρόοδο ή όχι και να δούμε τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν. Πέρα από αυτά υπάρχει βέβαια και ο προσδιορισμός του τι θέλουμε να πετύχουμε. Στα τέλη του Ιουνίου θα υπάρξει το τελικό κείμενο και να ξέρετε ότι έχει προετοιμαστεί σε συνεργασία με τη διαδικασία του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ό,τι εντοπίστηκε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ταιριάζει με τα όσα έχει εντοπίσει ω ανάγκε το ΝΑΤΟ. Άρα και οι ικανότητε που θα προωθήσουμε μέσω των μηχανισμών αυτών που σα περιέγραψα πριν εξυπηρετούν συγχρόνω και του σκοπού και του στόχου του ΝΑΤΟ. Συνεπώ, οι αμυντικέ ικανότητε, ωραία, αν ήταν μόνο αυτό, έτσι κι θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Και αυτό μόνο να ήταν. Αλλά έχουμε προχωρήσει πιο πέρα. Έχουμε δει τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε στα ανατολικά μας, νότια. Και υπάρχει ένα στοιχείο κλειδί εδώ. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιε προκλήσεις, χρειαζόμαστε κινητικότητα. Πρέπει οι δυνάμει μα να μπορούν να μετακινούνται. Και εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με κοινέ προσπάθειες ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η στρατιωτική κινητικότητα. Εσεί, κάπως αλλιώ το λέτε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Α, και εσεί έτσι το λέτε. Α, ωραία. Έχουμε την ίδια ορολογία λοιπόν. Αλλά κάπου είχα διαβάσει κάτι διαφορετικό, μια άλλη διατύπωση. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου, δεν την ακούμε. Ωραία. Στρατιωτική κινητικότητα λέτε. Καλώς. Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά προγράμματα στη συνεργασία ευρωπαικη Ευρωπαϊκή ΝΑΤΟ. Και εδώ τι κάνουμε. Η Ευρώπη εδώ μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο για ανάπτυξη υποδομών μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε με ρυθμιστικά διαδικαστικά ζητήματα, απλοποιώντας τις ελληνικές διαδικασίες, μεταφορά επικίνδυνων ε, αγαθών για στρατιωτικούς σκοπούς, αντιμετώπιση απειλών κλπ. κλπ. Δηλαδή εδώ υπάρχουν ένα σωρό προσπάθειε που μπορούν να γίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τη στρατιωτική κινητικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και το ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό και προσπαθούμε να δούμε όχι μόνο το εξαιρετικό έργο του ΝΑΤΟ, όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα, αλλά προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε και στους δικούς μας στους στόχους, αλλά να ικανοποιήσουμε και τις στρατιωτικέ απαιτήσει που θα προσδιοριστούν κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη του μήνα και θα εγκριθούν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Οπότε, στρατιωτική κινητικότητα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί πάνω στο οποίο συνεργαζόμαστε, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο. Μιλάμε για τα ίδια απειλών που αντιμετωπίζουμε. Οι υβριδικέ απειλέ είναι κάτι που έχουμε εντοπίσει εδώ και μερικά χρόνια και πάνω σε αυτό πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο. Και μάλιστα από τις 74 δράσεις, οι 20 έχουν να κάνουν με υβριδικέ ακριβώς απειλέ. Διάφορε δράσεις έχουν αναλυθεί. Υπάρχει ένα κέντρο αριστείας στο Ελσίνκι όπου συνεργαζόμαστε και ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανταλλάσσουν ιδέες. Επιπλέον όμως έχουμε φτιάξει και έναν πυρήνα υβριδικών απειλών επίσης που, ε, όπου συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ και καταλήγουμε σε κοινέ. Μάλλον, συγγνώμη, όχι κοινέ, συντονισμένε αναλύσει. Αυτή είναι η σωστή ορολογία για τις οποίες ενημερώνουμε τις χώρες μέλη. Είναι σωστό λοιπόν ο εντοπισμός των υβριδικών αυτών απειλών. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά. Μπορούμε να συνεργαστούμε λοιπόν για να εντοπίσουμε, να δούμε από πού προέρχονται και στη συνέχεια να τις καταπολεμήσουμε. Όχι μόνο να βρούμε από πού προέρχονται. Σε αυτό επίσης λοιπόν συνεργαζόμαστε. Τώρα για να καταλάβουμε καλύτερα την φύση των απειλών αυτών έχουμε ενισχύσει την συνεργασία μας και σε ασκήσεις. Ήδη πέρυσι είχαμε την πρώτη συντονισμένη και παράλληλη τέτοια άσκηση με βοήθεια στον ΝΑΤΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτο θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Ήταν τον Νοέμβριο προηγούμενη φορά. Τώρα θα ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για κινητοποίηση ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. 15 γενικοί διευθυντέ τη Κομισιόν κινητοποιούνται από έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο με θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, τις μεταφορές, την ενέργεια. Άρα κινητοποιείται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δικό μας μέσο αντιμετώπισης κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βασιζόμαστε σε ένα σενάριο υβριδικό και θα υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με τις κυβερνοαπειλές που ξέρετε ότι είναι και αυτές πολύ σημαντικέ απειλέ που έχουμε τελευταία. Η κύρια άσκηση λοιπόν θα είναι υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με από το ΝΑΤΟ. Έτσι θα κατανοήσουμε καλύτερα πώς αντιδρούμε στις απειλές αυτές και πώς μπορούμε μαζί να αντιδράσουμε σε αυτές τις απειλές αλλά παιδεία είναι οικοδόμηση ικανοτήτων. Πάλι συνεργαζόμαστε σε χώρες ε, πειραματικά, είτε είναι Μολδαβία, είτε είναι Ισία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, αλλά και σε άλλες χώρες, Ουκρανία, Γεωργία, Ιορδανία και κοιτάμε να δούμε μάλιστα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί για να βοηθήσουμε στο Ιράκ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ε, χώρες και περιοχές όπου δραστηριοποιούμεθα. Ε, Νότια Μεσόγειος, υπάρχει το Σιγάρι, υπάρχει το Σόφια και προσπαθούμε να δούμε και πού αλλού θα μπορούσαμε να δράσουμε μαζί όσον αφορά θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Άλλοι τομείς, οριζόντια τώρα, που καλύπτουν όλες τις ε, δραστηριότητές μας, είναι ε, γυναίκες, ειρήνη. Θα έχουμε ένα πρώτο εργαστήριο με ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό, γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια, το Σεπτέμβριο. Και τέλος να αναφερθώ και στην αντιτρομοκρατία, γιατί οι περισσότερες απειλές έχουν να κάνουν και με την τρομοκρατία. Είχαμε ένα πρώτο διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδο προσωπικού και επικεντρωθήκαμε στη συνεργασία για να υπάρξει αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών, πώς θα ε, κερδίσουμε το ISIS κλπ. Τα περισσότερα από αυτά θα υπάρχουν στην τρίτη έκθεση πρόοδου. που είναι η συνέχεια της Βαρσοβίας και θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα. Οι χώρες μέλη θα μας δώσουν κατευθυντήριες γραμμές και από πλευράς ΝΑΤΟ και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη αυτή τη βδομάδα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου προσβλέπουμε και σε παρετέρω εξελίξει όσον αφορά αυτή τη σχέση, όχι με παραπάνω δράσεις, αλλά με την υλοποίηση των όσων ήδη έχουμε αποφασίσει, που είναι ήδη πολλά. Ελπίζουμε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την διάσκεψη του ΝΑΤΟ του Ιουλίου να έχουμε μια νέα κοινή δήλωση με τους δύο προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής αλλά και του ΝΑΤΟ κάτι το οποίο θα μας δώσει νέα όθηση σε αυτήν την τόσο σημαντική σχέση και συνεργασία. Θα αναγνωρίζει τη σημασία των όσων ήδη από κοινού κάνουμε και θα δίνει και νέα, όθηση σε αυτές τις κοινέ προσπάθειες. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Εννοείται ότι όλα αυτά τα κάνουμε σεβόμενοι τις ε, διάφορες αρχές, διαφάνεια, αυτονομία των αποφάσεων και των διαδικασιών, συμμετοχή όλων, αμοιβαιότητα και ασφάλεια για όλους. Και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω και να συμμετάσχω σε αυτή τη συνάντηση και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Rose για τη συνεργασία μας. Επιβεβαιώνω ότι είπα ότι εκπρόσωπος και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να συνεχιστούν αυτοί οι κοινοί στόχοι. Μας δώσατε λοιπόν πολλές πληροφορίες. Uh, Δεν γίνεται αυτό συνήθως, αλλά φυσικά θα αποτελέσει και το έναυσμα για πολλές ερωτήσεις μετά ε, το καλωσόρισμα στην επόμενη ομιλήτρια μας, την κυρία Γκιότερ Μίλλερ, αναπληρωτή Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ, πρώτη γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Συγχαρητήρια λοιπόν και για ε, το γεγονός ότι είστε μια εξαιρετική διπλωμάτης, αλλά και προωθείτε την ε, εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Υπάρχει εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη και πολύ καλή εμπειρία σε ενεργειακή διπλωματία, αν μου επιτρέπετε να το πω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και εις βάθος τι συμβαίνει σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Να σας δώσω λοιπόν απευθείας το λόγο, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όλοι εκτιμούν την παρουσία σας εδώ και θα υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις ε, προς εσάς. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι εξαιρετική ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ σήμερα και μου δίνετε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ στο ίδιο βήμα με τον ε, σύντροφό μου στα όπλα, τον Παύλο Σεράνο. Κάνουμε αρκετή δουλειά μαζί. Ο Πέντρο έκανε εξαιρετική δουλειά, αναφέρθηκε στι λεπτομέρειε τη συνεργασία μα ε, στι ε, κομβικέ στιγμές και επομένω απλώ θα κάνω κάποιε προσθήκε. και πιστεύω ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσετε και τα σχέδιά μα για τη σύνοδο για τον άτομο που θα γίνει στα μέσα Ιουλίου και τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθούμε εκεί πέραν του θέματος ε, της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κάνω και τα δύο. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ε, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Πέντρο για την εξαιρετική συνεργασία και το γεγονός ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την εξαιρετική και ταλαντούχα ομάδα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους οποίους είμαστε σε επαφή καθημερινά με το προσωπικό μας ε, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ ε, και πιστεύω ότι υπάρχει πλέον ένα συνδετικό ιστός μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε μετά από την κοινή δήλωση στη Βαρσοβία και τις περιβόητες 84 προτάσεις, οι οποίες πλέον έχουν περάσει στο στάδιο της εφαρμογής και μάλιστα ε, κάποιες από αυτές είναι στην ενεργό υλοποίηση. Ε, είναι λοιπόν πολύ παραγωγική και αυτή η συνεργασία και ελπίζω να συνεχιστεί. Να σας πω και δύο λόγια στην αρχή για να σας παρουσιάσω λίγο και την προοπτική του ΝΑΤΟ για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Καταρχήν, και αναφέρθηκε και ο Πέντρος αυτό, οι δύο οργανώσεις μας αντιμετωπίζουν κοινέ προσκλήσεις ασφαλείας. Και οι δύο είναι πολύ αποτελεσματικές ε, στην ανταπόκριση αυτών των προκλήσεων από κοινού. Το 94% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλωστε ζει σε μια χώρα του ΝΑΤΟ. Επομένως έχουμε κοινέ προκλήσεις. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο καταλαβαίνουμε ε, εν γενός, είναι ότι ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτουν όλα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις ε, προκλήσεις ασφαλείας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά πιστεύουμε ότι μαζί έχουμε μια πλήρη εργαλειοθήκη και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Η δήλωση του Συνόδου της Βαρσοβίας ε, ζήτησε νέα όθηση και να προσδώσει νέα ουσία στη στρατηγική σχέση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε έχει γίνει πρόοδος άνευ προηγουμένου για να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία και δεν θα σας πω και πάλι τα πολλά κοινά προγράμματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πέδρο, αλλά θα ήθελα απλώς ε, να συμφωνήσω με την ουσία και τις προτεραιότητες ε, που τόνισε στις παρατηρήσεις του. Θα ήθελα κυρίως ε, να χαιρετήσω το έργο μας ε, για τις ε, προκλήσεις ε, για την κυβερνοασφάλεια και κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα, τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια, κάτι το οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε ε, και θα μας ασχολήσει ιδιαίτερα την επόμενη περίοδο. Ε, επίσης, θα ήθελα να τονίσω και το γεγονός ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει και η κοινοβουλευτική κοινότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόλις είπε ο Γενικός Γραμματέας την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, πριν από μία εβδομάδα ακριβώ στη Βαρσοβία ε, είχαμε συνάντηση της κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης του ΝΑΤΟ και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Στόλτεμπεργκ, αναφέρθηκε σε αυτό εκεί. Επίσης ε, το τόνισε σε πολλές ε, φορές ε, που έχει έρθει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Υποεπιτροπή Άμενας. Να σας πω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα που ενημερώνουμε τις επιτροπές σας από καιρούς καιρών και χαιρόμαστε που έτσι υπάρχει μια επικοινωνία και εταιρική σχέση. Η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει περαιτέρω δυνατότητες για συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ και το εκτιμούμε ιδιαίτερως. Τώρα, ο Γιάννη Στόλεμπεργκ πολύ συχνά τονίζει δημοσίω και ότι υποστηρίζουμε ε, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ε, άμυνας και πιστεύουμε ότι η ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα είναι πολύ καλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη και για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Συνεισφέρει σε περισσότερη κατανομή βαρών που όπως ξέρετε ήταν και φλέγον θέμα, θα το αναφέρω και αργότερα, αλλά ενισχύει και τον διατλαντικό σύνδεσμο, πιστεύουμε. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία τονίζουμε και ο Γενικό Γραμματέα τόνισε αυτέ τι τρει αρχέ, όπω τι αποκαλεί, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Καταρχά, ότι μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμπληρώσει και όχι να επικαλύψει τι προσπάθειε του ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι η άποψη που ε, έχουν εκφράσει σαφώ και οι Ευρωπαίοι ηγέτε. Επομένω, δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με απόψει οι οποίε εκφράζονται τα διάφορα κράτη, όπως το βλέπουμε, θα έχουν ανταγωνιστικές ε, Στρατιωτικέ απαιτήσει και φυσικά θα πρέπει να συμπληρώνονται όλο αυτό. Επίση, οι δυνάμει και οι ικανότητε που αναπτύσσονται από τι ευρωπαϊκέ ε, πρωτοβουλίε, θα πρέπει να δανείζονται στο ΝΑΤΟ αν υπάρξει ανάγκη. Χώρε που ανήκουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν και το περιθώριο να έχουν δύο ομάδε δυνάμεων και ικανοτήτων που να χρησιμοποιούνται ξεχωριστό, σε ξεχωριστό πλαίσιο. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη ε, αυτό όσο προχωρούμε. Και τέλο, ε, μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα λένε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ε, συμμάχους ε, του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμενοι βέβαια πάντα την αυτονομία και την ακαιρεότητα του κάθε οργανισμού και εδώ θα ήθελα να τονίσω και την αυτονομία και ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σαφώς ε, διακριτή και αυτό το αναγνωρίζουμε. Κάτι περαιτέρω τώρα γι' αυτό ο Γέντς ε, το τονίζει αυτό και ίσως πρέπει να επιστήσω και την προσοχή σας στο γεγονός αυτό. Το ΝΑΤΟ έχει μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια συνεχίζουν να δεσμεύονται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδάς αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία εδώ στην Ευρώπη και νομίζω ότι θα μάθετε περισσότερα γι' αυτό στο πλαίσια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στα μέσα του Ιουλίου. Μετά από το Brexit, ε, οι μη Ευρωπαίοι εταίροι θα είναι το 80% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ και τρεις από τις τέσσερις ομάδες μάχης ε, ε, θα έχουν στην ηγεσία του Σ ε, ε, συμμάχου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένε Πολιτείε, τον Καναδά και μετά τον Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Τώρα, να πω δύο λόγια παραπάνω για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου θα υπάρχει η συνεργασία ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο επίκεντρο. Ε, θα είναι από τα βασικά στοιχεία. Ο Γενικός Γραμματέας ο Στόλτεμπερκ και ο πρόεδρος Τούσκ και ε, ο πρόεδρος Γιούνκερ σκοπεύουν να υπογράψουν ε, μία δήλωση για να επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνοπτική έκθεση για την εφαρμογή των 74 προτάσεων θα δημοσιευθεί εντός ολίγου όπως είπε ο Πέτρο και θα δείξει ότι έχει γίνει πολλή δουλειά αλλά εκρεμούν ακόμα πάρα πολλά. Θα υπάρξει λοιπόν μια νέα κοινή δήλωση για να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει αυτή η συνεργασία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από αυτή την προοπτική. Τώρα, όσον αφορά τη σύνοδο αυτή καθ' αυτή, το βασικό στοιχείο θα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε, διότι τα θέματα αποτροπής και άμυνας ε, δεν αφορούν μόνο τις δυνάμεις που έχουμε αναπτύξει στις τέσσερις ομάδες μάχης ε, ε, στα κράτη της Βαλτικής και στην Πολωνία, αλλά επίσης και στη δυνατότητά μας να κινητοποιήσουμε δυνάμεις και να τις ενισχύσουμε γρήγορα αν χρειαστεί. Αυτό σχετίζεται με τη σειρά του, με την ετοιμότητα των δυνάμεών μας και τις δυνατότητες να μετακινήσουμε και δυνάμεις ε, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Έτσι μπορούμε να έχουμε αποφάσει όσον αφορά την ενίσχυση, την ετοιμότητα και τη στρατιωτική κινητικότητα, όχι μόνο πέρα του Ατλαντικού, αλλά και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μάθετε και λίγα περισσότερα γι' αυτό από το Γενικά Διευθυντή του τον επιτηλά έρχη μάλλον του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα είναι εδώ στο επόμενο ε, πάνελ και θα σας ε, ε, πει πολλά πράγματα, είναι η Δήμον επί του θέματος. Ε, εγώ μπορώ να απαντήσω ότι θέλετε, αλλά ο Γιάννη είναι αυτός ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Η Ρωσία φυσικά θα συμπεριλαμβάνεται στις συζητήσεις μας. Υποθέτω ότι οι ηγέτες θα θέλουν να τονίσουν ότι το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει μια διτή προσέγγιση από τη Σύνοδο της Βαρσοβίας και μετά όσον αφορά τη Ρωσία, που αφορά την αποτροπή και την άμυνα αφενός και τον πολιτικό διάλογο αφετέρου η αποτροπή και άμυνα για να στείλουμε στη Ρωσία ε, συνεχώς ένα ισχυρό μήνυμα και αποφασιστικό μήνυμα ότι όποτε παρουσιάζουν διεθνέ δίκαιο και διεθνεί κανόνες θα λαμβάνουν και μια αποφασιστική απάντηση από πλευράς ε, συμμαχία Διάλογο, διότι πρέπει να διαχειριστούμε και τη σχέση μας με τη Ρωσία και να προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε αν μπορούμε. Ασχολούμαστε λοιπόν με τα θέματα του διαλόγου. Την περασμένη Πέμπτη έγινε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Ρωσία ε, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ και πιστεύουμε ότι ο διάλογο ε, συμβάλλει σε περισσότερη προβλεψιμότητα στη σχέση μα με τη Ρωσία και ελπίζουμε και αμοιβαία ασφάλεια σιγά σιγά και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ίσω και προβλήματα τα οποία αναδύθηκαν κυρίω όσον αφορά στρατιωτικά ατυχήματα και περιστατικά τα οποία ε, κατά πάσα πιθανότητα θα συμβούν πιο συχνά λόγω και αριθμού των δραστηριοτήτων σε περιοχέ στι οποίε η συμμαχία του ΝΑΤΟ ε, έρχεται αντιμέτωπη με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η προστασία της σταθερότητας αφορά και την ε, προστασία της σταθερότητας στη γειτονική μας περιοχή, γιατί όταν είναι σταθερή οι γειτονέ μας είμαστε πιο ασφαλείς. Και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει πολλούς ε, γείτονες, και ο καθένα έχει τις δικές του μοναδικές συνθήκες. Η Ουκρανία, η Γεωργία, τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ορδανία, η Τινησία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και πολλές άλλες χώρες τι οποίες δραστηριοποιείται το ΝΑΤΟ. Το ε, προωθεί την σταθερότητα με διάφορα μέσα, από εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων, δημιουργία ικανοτήτων, πρακτική και πολιτική στήριξη. Αλλά αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός τομέας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που ο Πέντρο τόνισε και την πιλωτική μας δραστηριότητα με χώρες όπως για παράδειγμα η Ορδανία και η Τινησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και καλωσορίζω και το πιλωτικό πρόγραμμα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η συζήτηση για τον εξυγχρονισμό στη Σύνοδο θα τονίζει και το γεγονό ότι το περιβάλλον ασφαλείας είναι μεγαλύτερη πρόκληση τώρα από το τέλο του ψυχρού πολέμου και μετά. Το ΝΕΤΟ πρέπει να αναβαθμίσει τι προσπάθειε του για να αντιμετωπίσει τι προσκλήσει και να προσαρμοστεί ταυτόχρονα. Ελπίζω λοιπόν οι ηγέτε να εγκρίνουν και αλλαγέ στι δικαιτικές δομέ του ΝΑΤΟ και αυτό φυσικά θα έχουμε και μια ατλαντικό, ένα ατλαντικό στρατηγείο στο Νόρφολκ στη Βιρτζίνια και ένα τμήμα ε, επιμελητίας ε, στήριξης το οποίο θα φιλοξενείται στη Γερμανία. Ταυτόχρονα ε, γίνεται μετατροπή του στρατηγίου του ΝΑΤΟ, ώστε να είμαστε διάφανος, ευέλικτος, αποτελεσματικός μηχανισμός. Και αν δείτε και το νέο μου σχεδιασμό, θα δείτε ότι θέλουμε να είμαστε διάφανοι εκφύσεων. Και Μόλις μπήκα σε αυτό το όμορφο κτίριο, διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες ε, ε, με τη βασική είσοδο και ε, την κεντρική είσοδο στην στο κτίριο, αλλά θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα της διαφάνειας στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και τη ασφάλειας ταυτόχρονα. Και τέλος, ε, κάτι βεβαίως ε, εξίσου σημαντικό, κατανομή βαρών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στη Washington αυτή τη στιγμή, ε, στο επίκεντρο της παρούσας κυβέρνησης στη Washington, αλλά φυσικά και εμείς έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τις δαπάνες, ε, θέλουμε να ε, καλύψουμε την ε, δέσμευση να δαπανάτε το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα. Ο Πέδρο υπενθύμησε ότι το συμφώνησαν οι σύμμαχοι πριν από δύο χρόνια. Στην πραγματικότητα το συμφώνησαν πριν από τέσσερα στην Σύνοδο της Ουαλίας το 2014. Αλλά αφορά και συμβολή σε αποστολές του ΝΑΤΟ και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να παρέχονται οι απαραίτητες δυνατότητες και ικανότητες στη συμμαχία. Ε, υπάρχουν επίσης θετικά νέα για πολλές ε, δυνατότητες ε, και επίτευξη στόχων. Για παράδειγμα, το 2004 μόνο τρει σύμμαχοι δαπανούσαν το 2% του ΑΕΠ του στην άμυνα. Φέτος επιτρε... Ε, περιμένουμε 8 χώρες, ε, με περισσότερες χώρες να οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό φυσικά θα είναι και πρωτεύον ζήτημα στις συζητήσει ε, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και φυσικά προσβλέπουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορμή που θα λάβουμε από τη Σύνοδο των Βρυξελών για την επόμενη χρονιά, γιατί το 2019 είναι η 70η επέτειο της συμμαχίας, είναι στρατηγική σημασία χρονιάς λοιπόν για το ΝΑΤΟ για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους βασικούς βασικούς στόχους ε, και να δούμε πώς θα περάσουμε στην επόμενη περίοδο, στην επόμενη δεκαετία και θεωρούμε ότι θα είναι και εφαλτήριο για ε, ε, να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα και αυτό θα μας το βοηθήσει να το κάνουμε και η Σύνοδος των Βρυξελών τον Ιούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε σήμερα. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία και προσβλέπω στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Well, thank you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτιμούμε πάρα πολύ το χρόνο σας, ε, το ότι ήρθατε εδώ για να ενημερώσετε τα μέλη για την ε, κατάσταση και τις προοπτικές της ε, συνεργασίας μας. Νομίζω πως έχουν μαζευτεί αρκετές ερωτήσεις, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όποιον έχει κάποια ερώτηση, όποιο από τα μέλη θα ήθελε. Θα ήθελα να δω πρώτα ποιος επιθυμεί να πάρει το λόγο. Νομίζω πως ε, ξεκινήσατε ε, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ένα συνάδελφος από την Πορτογαλία, ο κύριος Μιράντα Καλία. Δεν σας βλέπω καλά, αλλά έχετε το λόγο. Θα γίνουν πρώτα δύο-τρει ερωτήσει και ύστερα θα δώσουμε το λόγο στου καλεσμένου. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και την θετική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα δύο τελευταία χρόνια που πλησιάζει η Σύνοδο ε, Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και θεωρώ πω πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό για να, να επικεντρωθούμε πιο φιλόδοξα στην συνεργασία. Εσείς ε, πώς βλέπετε τα πράγματα και έπειτα κατά τη διάρκεια της συνόδου θα εγκριθεί από τη συμμαχία, θα εγκριθεί από τη συμμαχία ένα ε, κείμενο. Ε, επίσης, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δράσεις για την ε, ασφάλεια. Τι γίνεται λοιπόν για την ανάπτυξη δυνατοτήτων των ε, χωρών εταίρων και για την αύξηση της δικής τους ανθεκτικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις, αν δεν σας πειράζει. Εσείς, ο συνάδελφο από τη Λετωνία. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές. Βέβαια, να πω πως ε, στη Λετωνία στηρίζουμε και τους διοργανισμούς, διότι είναι αναγκαίοι για την ύπαρξή μας και για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λοιπόν αναγκαία η συνεργασία. Όταν γίνεται λόγος για νέες απειλές, ε, να πούμε ότι μία από αυτές είναι και εσωτερική απειλή. Ο εξτρεμισμός, ο λαϊκισμός είναι κάτι που έχει πολιτική χρειά και αυξάνει την ε, απειλή που ασκούν εξωτερικές δυνάμεις επίσης. Όπως είπατε κι εσείς, γίνονται προσπάθειες και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει το κέντρο αριστεία στο Ελσίνκι για τον υβριδικό πόλεμο, αλλά υπάρχει και στη Ρήγα ένα ερευνητικό κέντρο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εσάς ε, σε ποιο βαθμό συνεργάζονται αυτοί οι δύο οργανισμοί και ποιες είναι οι διαφορές σε αυτά που κάνουν. Διότι προσπαθούμε με να αντιμετωπίσουμε την εσωτερική απειλή που απειλεί περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που αφορά λοιπόν περισσότερο εμάς. Όμω, όπως γνωρίζετε, του χρόνου έχουμε ευρωεκλογέ. Και κάθε μήνα στην Ευρώπη διεξάγονται εκλογές και βλέπουμε όλο ένα και αυξανόμενα αντιευρωπαϊκά και αντινατοϊκά συναισθήματα. Ε, που εκπροσωπούνται εν μέρει και από κυβερνήσεις που είναι δημοκρατικά εκλεγμένες παρότι τα επιχειρήματά τους δεν είναι και τόσο ε, πολιτικά ορθά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τάνοκ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκ μέρου του Ηνωμένου Βασιλείου. Είστε λοιπόν ε, μπαλαντέρ και στα δύο όργανα. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, τους προσκεκλημένους να πω πως είμαι σχεδόν 20 χρόνια ευρωβουλευτής, ασχολούμαι με αυτά τα θέματα και παρότι είμαι συντηρητικός είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι μειοψηφία στη χώρα μου δηλαδή. Ένας ομιλητής αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία στα 80% των δαπανών στο ΝΑΤΟ οι οποίες θα, οι οποίες θα γίνονται από μη ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφού... αφού το αποχωρεί στο Ηνωμένο Βασιλείο από αυτή. Δεν ξέρω αν είναι αυτό απειλή, πάντως σίγουρα θα αποτελέσει πρόκληση στη νέα πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όμως ε, σίγουρα θα υπάρξει σημαντικό κενό στον προπολογισμό, 15 περίπου δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω εάν οι άλλοι μεγάλοι συνεισφέροντε, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, ε, θα είναι διατεθειμένες να καλύψουν αυτό το κενό. Υπάρχουν λοιπόν ε, διάφορες πρωτοβουλίε που ελπίζω ότι δεν θα επηρεαστούν από την αποχώρηση της χώρα μου. Διάφορα προγράμματα, διάφορα ταμεία όπω το Ταμείο ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Χρειάζεται λοιπόν μια κάποια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη και την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση των πραγμάτων. Ας μην ξεχνάμε βέβαια και την ανακοίνωση Τραμπ για του τιμωρητικούς δασμούς ε, στις εξαγωγές σε χάλιβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, σε αυτές τις εξαγωγές συμπεριλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινά εμπορικό πόλεμο και αυτό που μας εκπλήσει δεν είναι τόσο αυτό, αλλά ότι αυτοί οι δημορτικοί δασμοί επεκτείνονται και ε, επηρεάζουν και τον Καναδά. υπήρξαν δρυμίες ε, κριτικές και από το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα δεδομένου ότι μέχρι τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ο κυριότερος σύμμαχός μας. Οι εξελίξεις λοιπόν είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, αρκετά περίεργες θα έλεγα και νομίζω πως όλες οι παρεμβάσεις το τόνισαν. Μάλιστα, νομίζω πως ε, αρκούν οι ερωτήσεις, ιδιαίτερα μετά από την τελευταία, γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Κότε Μόλερ. Σας ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, περισσότερο σχόλια ήταν αυτά που ακούσαμε παρά ερωτήσεις. Ε, θα σταθώ όμως αυτό που είπατε ότι συμβαίνουν διάφορα περίεργα αυτόν τον καιρό. η τιμωρητική δασμή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται και έτυχε το Σαββατοκύριακο να παραβρεθώ στη Σιγκαπούρη, στο συνέδριο, σαν γκριλιά που ακούστηκαν αυτά τα σχόλια για τους ε, τιμωρητικούς αυτούς δασμούς. Υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για αυτόν τον ε, πόλεμο που χρησιμοποιεί τους δασμούς και νομίζω πως θα αποτελέσει μεγάλο και σημαντικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα βέβαια αυτά και νομίζω πως ε, ο τρόπος που έχουν προσεγγιστεί θα οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν πως ε, όσα ακούστηκαν στο Σαγκριλέ ήταν αρκετά σημαντικά και είχα την εντύπωση πως ε, εστάλει ένα μήνυμα ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για συζήτηση. Τώρα, να απαντήσω στον συνάδελφο από την Πορτογαλία, ο οποίος ρώτησε για τις διάφορες δυνατότητες ε, συνεργασίας και ανάπτυξη αυτής. Νομίζω πως μέρος αυτής της συνεργασίας προέρχεται από τις ε, διάφορες ευθύνες, καθημερινές ευθύνες που έχουμε και οι δύο. Βέβαια είναι και ζήτημα ανθρώπινων πόρων. Ε, τι χρειάζεται από πλευράς ανθρώπινων πόρων για να συνεχίσουμε, για να μπορούμε να ε, υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας. Νομίζω λοιπόν πως εδώ έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος και στα έργα και τα προγράμματα που ανέφερε ο Πέντρο και πιστεύω πως ε, πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, Σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη προσοχή το θέμα των διαθέσιμων πόρων έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, αναβολές και καθυστερήσεις ε, στα διάφορα προγράμματα και πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόοδος. Διότι ο καιρός περνά. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε πως πρέπει να διασφαλιστεί το ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας σε βάση των τριών ε, κυριότερων αρχών. Θα τις επαναλάβω στη συνέχεια, όμως να τονίσω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αρχές που θεωρώ πως θα πρέπει να συνεχίσουν να διέπουν τη συνεργασία μας. Διότι από αυτές θα εξαρτηθεί και η πρόοδος ε, που θα σημειωθεί. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, όπως είπα και νωρίτερα, πως ε, σίγουρα είναι πολύ σημαντική η προβολή της σταθερότητας. Σίγουρα δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν άλλα προγράμματα, όμως η σταθερότητα και η προβολή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πιστεύω πως αυτή είναι, αυτό είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρώσουμε και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη κάνουν αρκετές ενέργειες πάνω σε αυτό. Και θεωρώ πως στο ΝΑΤΟ θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας, το είπα και ευθύ εξ αρχής κιόλας, μόνο εάν χρησιμοποιήσουμε όλα τα ε, διαθέσιμα εργαλεία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί. Και θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι η οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία είναι το μίσο που το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία ανάμεξη. Γι' αυτό ε, η συνεργασία σίγουρα θα εξαρτηθεί και από τις σχέσεις που έχουμε με τους εταίρους ε, στο νότο της Συμμαχίας και στη Μέση Ανατολή. Είναι λοιπόν εκ των όνου αυτή η σωστή και καλή συνεργασία με τους εταίρους μας. Χρειάζεται συνεργασία στην ανάπτυξη δυνατοτήτων, ε, υποδομών, στον τομέα της ασφάλειας γενικότερα. Όμως υπάρχουν και άλλοι τομείς συνεργασίας. Υπάρχει η οικονομική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ επίσης που βλέπω εδώ τον συνάδελφο από τη Λετωνία. Τελευταία φορά νομίζω τα είπαμε στη Ρήγα σε ό,τι αφορά αυτά που είπατε, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε στις ασύμετρες ή υβριδικές απειλές. Και στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ σημαντικές συζητήσεις σε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του ανώτατου οργάνου μας δηλαδή, για θέματα τα οποία είναι υψίστον ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προχωρήσουμε στηριζόμενοι πάνω στην δημιουργία γνώσεων, συλλογή πληροφοριών και γι' αυτό λοιπόν το Κέντρο Εκμετώπισης Ευρυθικών Απειλών στο Ελσίνκι μας βοηθά να κατανοήσουμε την ουσία του προβλήματος. Διότι οι απειλές αυτές που είναι απειλές ε, σε πολλές κατευθύνσεις και ε, στο εκλογικό μας σώμα, τους ψηφοφόρους μας, είναι κάτι που δεν μπορούμε να παραμελήσουμε. Χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό και να καταφέρουμε να ελέγξουμε τις απειλές αυτές. Το Φεβρουάριο που πήγα στη Ρήγα επίσης, να πω ότι ότι εξεπλάγει με την πρόοδο που σημειώνεται εκεί και σίγουρα πρέπει εμείς να προλάβουμε αυτές τις επιθέσεις στη δημοκρατία μας. Υπήρξαν ε, προτάσεις τις οποίες θεωρώ πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουμε. Δεν ξέρω τι θα ήθελε να πει και ο Πέντρο πάνω σε αυτό, όμως νομίζω πως η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών προχωρά με καλούς ρυθμούς. Έγινε μια κίνηση πέρυσι, ε, αλλά τόσο τα κέντρα στη Ρήγα όσο και στο Ελσίνκι νομίζω πως κάνουν εξαιρετική δουλειά. Πέντρο Σεράνο, ναι, εσύ τώρα. Η σειρά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συμφωνώ περίπου με όλα όσα είπε η αναπληρώτρια Γενικός Γραμματέας Όλος Παραδόξος. Το Όλος Παραδόξος ε, το λέω βέβαια χαριτολογώντας γιατί προφανώς και συμφωνούμε για το Brexit και για το ότι δεν συζητήσαμε γι' αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο το ξεκαθάρισε και πιστεύουμε ότι έτσι είναι πράγματι. Το Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν βγαίνει ούτε από την Ευρώπη, ούτε από την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη φυσικά. Το ότι δεν θα είναι χώρα μέλος δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει να συνεργάζεται σε θέματα Άμυνα και συνεργασία τώρα με τη μορφή που αυτά θα πάρουν και που δεν την ξέρουμε ακόμα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι για το συμφέρον και του Ηνωμένου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί ένας διακανονισμός προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Ξέρουμε πως έχει προχωρήσει η πολιτική άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν πάντα μια ανοιχτή πολιτική. Οπότε και αυτό όχι προ το δικό τη μόνο συμφέρον, αλλά για να προστατεύσει και άλλου. Οπότε πάντα πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία. Οπότε εφόσον η διαδικασία είναι ανοιχτή, υπάρχει πάντα περιθώριο να ε, καλωσορίσουμε στου κόλπου τη και άλλου, πόσο μάλλον μια χώρα που ανήκει στην οικογένειά μα μέχρι τώρα. Τώρα για τα πόδια και του περιορισμού. Υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες στον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα. Αυτά τα λέει και η ίδια συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζει το ρόλο του ΝΑΤΟ που είναι υπεύθυνο για την κοινή πολιτική των χωρών μελών του. Είναι σαφές αυτό. Και όλοι αρχίζουμε από αυτό το σημείο. Τώρα για τις τρεις κύριες αρχές στις οποίες αναφερθήκατε. Πολλές από αυτές είναι διαφυσβήτητες. Έχουμε ήδη πει ότι όλες οι ικανότητες που θα αναπτυχθούν δεν είναι παρά των χωρών μελών. Οπότε οι χώρες μέλη είναι που θα αποφασίσουν τι θα κάνουν για αυτέ τι ικανότητε όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε λοιπόν αναπτύσσεται στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να τι χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, σε συμμαχίε που έχουν ή οτιδήποτε άλλο. Για την μη επικάλυψη, για να είμαι ειλικρινή, το συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για την περιττή επικάλυψη, γιατί ίσως σε κάποιους τομείς να χρειάζεται κάποια ικανότητα ακριβώς που να διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αυτονομία για να προχωρήσει στη μία ή την άλλη δράση που θεωρεί αναγκαίο να προχωρήσει μόνη της. Αυτό δεν συγκρίνεται βέβαια με την αποστολή του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την ίδια αρμοδιότητα όπως το ΝΑΤΟ για την προστασία των μελών. Οι δράσεις επίσης είναι διαφορετικές τις οποίες προχωράμε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη συμμετοχή μη, μάλλον συμμάχων μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στις δικές μας δράσεις. Οπότε αυτές είναι αρχές που έτσι καλλιώς δεν είναι επίμαχες και σίγουρα δεν αποτελούν εμπόδιο στο κοινό μας έργο. Καθάλλου. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα για τη σημασία που έχει η συνεργασία μας και να μην αφήνουμε περιθώρια για παρεξηγήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους δύο οργανισμούς και για την ασφάλεια των πολιτών μας και εννοείται ότι το φροντίζουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να στείλουμε σαφή μηνύματα για το πώς συνεργαζόμαστε υπέρ του κοινού όφελους και των δύο οργανισμών. Ε, συμφωνώ με την Ροζ. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες μας και το βλέπω καθημερινά είναι η ανθρώπινη πόρη. Πώς θα υλοποιηθούν δηλαδή όλες αυτές οι δράσεις που έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας. Και εδώ είναι ένα καλό μέρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα πούμε αυτά, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για τον προπολογισμό μας και πώς θα υλοποιήσουμε όλα αυτά που πρέπει να υλοποιήσουμε δεν έχουμε αρκετούς πόρους σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ αλλά και γενικότερα σε τομείς όπου πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες. Τέλος, για τις υβριδικές απειλέ, όπως είπε και η Ρόζ, το κέντρο στο Ελσίνκι μόλις αρχίζει τώρα. Προσφέρει ένα ευρύ πλαίσιο το οποίο διευκολύνει ανταλλαγές μεταξύ πυρογνωμόνων. Είναι ένας χώρος δηλαδή όπου πραγματογνωμοσύνη συγκεντρώνεται και αναλύεται. Ένα από τα βασικά στοιχεία, όπως είπε και η Ροζ, είναι η πρόληψη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δραστηριοποιηθεί για το θέμα της αντοχής και έχουμε διάφορα εργαλεία. για να ενισχυθεί η αντοχή μας. Αλλά το βασικό για τα ευρετικά είναι η ανάλυση του τι συμβαίνει και να συνδέουμε όλες τις τελίτσες, όλα τα κομματάκια του παζλ για να διαπιστώσουμε κατά πόσο όντως υπάρχει απειλή, επίτηδες, να την εντοπίζουμε και δημόσια και να υιοθετούμε τα κατάλληλα μέτρα που μπορεί να είναι πολλά και διαφορετικά. Και αυτή είναι η δύναμη των διοργανισμών που όταν βάλουμε μαζί τις δυνατότητές μας μπορούμε να ανταποκριθούμε πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία. Και άλλες ερωτήσεις τώρα. Δύο-τρεις από σας. Ε, έχετε ερωτήσει. Μεσόγειος, Τουρκία. Παρακαλώ. Η ερώτησή μου, λίγο πολύ ρωτήθηκε από τον κύριο Κάνιτς, αλλά αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι το εξής. Όταν μιλάω για εσωτερικές απειλές, εγώ εννοώ κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που εννοεί εκείνος. Οπότε οι απαντήσεις σας δεν με ικανοποιούν. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μια διαφορετική οπτική γωνία. Ως εσωτερική απειλή ενώ θέματα όπως είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η ισλαμοφοβία, ο λακισμός. Τέτοιες απειλές έρχονται από την Ευρώπη αυτή καθευτή. Δεν πρόκειται για ευρυδικές απειλές ή άλλου είδους. Υπάρχει απόσταση όλο και μεγαλύτερη από τις βασικές αξίες που κανονικά είναι η ίδια η Ευρώπη. Και αυτό που θέλουμε να ονομάζουμε σήμερα Ευρώπη. Συνεπώς, αυτή η απόσταση από τις βασικές αρχές πιστεύω ότι αντί να είναι η Ευρώπη ένας ασφαλής λιμένας, γίνεται ένας καταστροφικός ε, χώρος. Ποια θα έπρεπε να είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα και τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την αποφυγή αυτών των ενδυνάμει εσωτερικών απειλών. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Θα στην Τουρκία ο κύριος Κονκάο. Έχει και αυτός μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, η ερώτησή μου είναι για την Ρόσ και το Μέλλερ. Είναι προφανές τώρα με αυτά που έγιναν στην Ουκρανία από πλευρά τη Ρωσία, ότι απελείται η ασφάλεια τη Ευρώπη. Για πρώτη φορά μετά το ψυχρό πόλεμο, η άμυνα, η αποτροπή, δυνατότητες δηλαδή άμυνας και αποτροπής ε, της Ευρώπης δοκιμάζονται από τη Ρωσία και τους ρωσικούς κανόνες. Και είναι ενισχυτικό που έχει ακολουθήσει υβριδικές τακτικές η Ρωσία που είναι πιο δύσκολο να εντοπίσει κανείς από ό,τι γινόταν παλιότερα παραδοσιακά. Θέλω να επιστήσω επίσης την προσοχή σας στην πυρηνική συνιστόσα της επιθετικής ρωσικής πολιτικής, διότι έχει μία ολοκληρωμένη πολιτική για συμβατικές ε, και πυρηνικές δράσεις, ασκήσεις και ξέρουμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια η πυρηνική συνιστόσα αποτροπής του ΝΑΤΟ ήταν στο περιθώριο. Δεν λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια ριζοσπαστική αλλαγή στην πυρηνική διάσταση στο ΝΑΤΟ εξαιτία αυτών των γεγονότων. Θα ήθελα όμως να ξέρω την άποψή σας για τις ικανότητες πολιτική, ε, πυρηνικής αποτροπής των συμμάχων και τι θα γινόταν εφόσον ε, μάλλον τι γίνεται εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει πυρηνική διάσταση στην ε, ρωσική στρατηγική. Έχουμε μετά και δύο ερωτήσεις, αλλά θα δώσω και στον Παύλο Άλε την ευκαιρία να υποβάλει και αυτό τις ερωτήσεις του. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την νότια πτέρυγα της Συμμαχίας και της Ευρώπης, που νομίζω ότι είναι ένα κοινό ζήτημα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε το μεταναστευτικό ε, πόσο πολύ επηρεάζει όχι μόνο την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, αλλά και την πολιτική κατάσταση γενικότερα στην Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και άλλες χώρες. Και δεν είναι μόνο θέμα της τρομοκρατίας, ε, είναι γενικότερα. Το ΝΑΤΟ, κατά τη γνώμη μου, πήρε μια σπουδαία απόφαση με τη στρατογική του ε, απόφαση αυτή η νέα δομή του ΝΑΤΟ πώς μπορεί να λειτουργήσει πλήρως, πότε και, πώς, και πότε θα μπορέσει να συνεργαστεί καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί από ό,τι κατάλαβα εγώ, στόχος της δομής αυτής δεν είναι τα στρατιωτικά ζητήματα, αλλά η κατανόηση των κανόνων που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο από την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται στην Αφρική. Οπότε, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών και, για παράδειγμα, κατάρτιση δυνάμεων στην Αφρική. Δεύτερον, Δυτικά Βαλκάνια. Είναι στην καρδιά της Ευρώπης και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έχουμε εδώ συναδέρφους από τη Σερβία, το Μαυροβούνι, που είναι πιο σταθερέ χώρε. Πάντως η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά το πώς βλέπουν τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπά αυτές τις χώρες. Τι πιστεύετε λοιπόν για την κατάσταση εκεί. Ιστορικά έχουμε δει πολλές χώρες στην περιοχή έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ πριν γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μπορεί να γίνει το αντίθετο στο μέλλον. Ποιο είναι το σχέδιο για τη συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Κύριε Γκέτεμελερ, νομίζω ότι έχετε αρκετές ερωτήσεις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, ναι, εξαιρετικές οι ερωτήσεις. για τους ε, Τούρκους συναδέλφους όσον αφορά το ρατσισμό, την ξενοφοβία. Ναι, είναι οι υβριδικές μέθοδοι, αν σας κατάλαβα καλά. Στο ΝΑΤΟ αρχίζουμε να προσπαθούμε να κάνουμε αναλυτικό έργο συνεχίζονται συζητήσεις και στη διάσκεψη, θα συνεχιστούν τον Ιούλιο. Και επικεντρωνόμαστε στις υβριδικές μεθόδους. Πιστέψτε με, δεν είναι κάτι καινούριο. Η μέθοδη υβριδικού πολέμου, όπως λέμε, είναι από τον νοτροϊκό Πόλεμο, έτσι, με το Δούριο Ήπο. Από την ε, τους αρχαίους χρόνους, λοιπόν, τον ξέρουμε το δόριο ύπο. Αλλά πρόκειται βέβαια και για την ε, διάλυση της ενότητας, για το πώς θα διχαστούν εταίροι, σύμμαχοι, προκειμένου να μην υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη, να υπονομεύεται αυτή και να υπονομεύεται και το σύστημα γενικότερα. Οπότε στο βαθμό που υπάρχουν προβλήματα σε πολλές κοινωνίες και στη δικιά μου χώρα και στις Ηνωμένε Πολιτείε, εδώ δεν έρχομαι ως Αμερικανίδα διπλωμάτης όπως ξέρετε, αλλά στέλεχος του ΝΑΤΟ, αλλά τα βλέπουμε αυτά τα προβλήματα. οι υβριτικοί μέθοδοι χρησιμοποιούνται ακριβώς για να μεγενθύνονται αυτά τα προβλήματα και ο στόχος τους είναι ο διχασμός μεταξύ κοινωνιών, χωρών, ώστε να επιδεινώνονται κάποιες τάσεις και να προκληθεί πραγματικά ζημιά στο κράτος δικαίου. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιου είδους απειλές. Και πράγματι θα μπορούσε κανείς να πει ότι μερικές φορές πρόκειται για προπαγάνδα που μπορεί να μην έχει αμέσως επιπτώσεις στρατιωτικές ή ασφάλειας, αλλά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπτώσεις στην ασφάλεια αργότερα. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλα αυτά. Μ' άρεσε έτσι όπως το περιγράψετε ότι απομακρυνόμαστε σταδιακά από τις αξίες μας. Πολύ καλά το θέτετε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να φροντίζουμε να υπάρχει συνδυτοποίηση όλο και περισσότερο, να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τέτοιες μεθόδους και στη Ρήγα το συζητήσαμε. Είπαμε να μην αφήνουμε τις θεωρίες συνωμοσία να κυκλοφορούν και να σπέρνουν ζυζάνια και να δημιουργούν ε, το φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Θα πρέπει από την αρχή να λέμε την αλήθεια και να αντιδρούμε όσο γίνεται πιο έγκαιρα. Δύσκολο βέβαια, γιατί σήμερα πώς να αντιμετωπίσει κανείς το βάρος αυτής προπαγάνδας με τόσους πόρους που διατίθενται μερικές φορές για αυτήν, για tweets και άλλες μεθόδους μηνυμάτων. Ε, Πολλέ ζητήματα δηλαδή τίθενται, αλλά το πρώτο είναι να κατανοήσουμε το πρόβλημα, να κατανοήσουμε την απειλή, να κατανοήσουμε τη μέθοδο που χρησιμοποιείται και μετά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σταματήσουμε και μετά να προλαμβάνουμε καταστάσεις όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο άμυνας, η αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Ψάχνουμε να βρούμε και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν έχω καμία τέλεια απάντηση αυτή τη στιγμή να σας δώσω, αλλά η συνειδητοποίηση υπάρχει, πρέπει να ξέρετε, και οι προσπάθειες γίνονται για την αντιμετώπιση. Κάτι όμως που θέλω να αναφέρω και το είπε και ο Πέδρο είναι η αντοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα πώς ε, θα αντισταθούμε στη, στο κυβερνοέγκλημα, στις κυβερνοπυλές αλλά υπάρχει και μία πτυχή της κοινωνίας που όντως αντέχει σε αυτή την παραπληροφόρηση. Πολύ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει δουλειά πάνω σε αυτά να καταφέρει να βρεθεί ακόμα πιο μπροστά, να προλαβαίνει τις καταστάσεις δηλαδή, γιατί η δουλειά που κάνει είναι πιο προθυμένη από αυτή που κάνει το ΝΑΤΟ από αυτού. Τώρα, χαίρομαι που σας βλέπω και εσάς. Τον Ιανουάριο είχαμε βρεθεί στην Τουρκία. Ξέρετε πώς έχω ασχοληθεί με τα πυρηνικά, την αποτροπή. Θα μπορούσα να μιλάω όλο το απόγευμα για αυτά τα ζητήματα. Δεν θα το κάνω όμως, να μην βαρεθείτε. Πάντως, η ικανότητα αποτροπής των πυρηνικών του ΝΑΤΟ ε, είναι σημαντική και πολλές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την ε, κατοχή της νέας γενιάς ε, πλατφόρμας είναι ικανότητε που θα επιτρέπουν στη χειρότερη περίπτωση να υπάρξει πυρηνική αποστολή. Βέβαια, αυτό είναι μέρος μόνο της όλης ιστορίας, γιατί υπάρχουν κέντρα αποτροπής που ασκούνται με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι τρεις πυρηνικές χώρες και κάθε μία από αυτές μέσα στο ΝΑΤΟ παίζει διαφορετικό ρόλο όσον αφορά την αποτροπή. Πάντως το πιο σημαντικό εδώ είναι να δούμε την αποτροπή σαν ένα ευρύ πρόβλημα γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και από πλευρά των υβριδικών απειλών που μας έρχονται, ασυμμετρικές απειλές. Μετά να δούμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που προβλέπει τι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση απειλής σε μια χώρα μέλος της συμμαχίας που θα ζητήσει βοήθεια. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι ήδη στη Βαρσοβία πριν από μερικά χρόνια είχαμε θεωρήσει και την κυβερνοαπειλή ότι εμπίπτει στα πλαίσια του άρθρου 5. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια εξέλιξη απειλών που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να αποτρέψουμε. Πάντως, όσον αφορά τα πυρηνικά, θεωρούμε την απειλή ε, μια πυρηνικής επίθεσης κάτι πολύ μακρινό. Φυσικά και πρέπει να παρακολουθούμε τις ικανότητες ε, όλων των ε, πλευρών, χωρών κλπ. Πάντως η πιθανότητα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρηνική επίθεση είναι κάτι πολύ μακρινό. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αλλά πρόκειται για όπλα και τονίζω ότι είναι, τα πυρηνικά όπλα είναι μαζικής καταστροφής. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, μεν, αλλά πρέπει να θεωρήσουμε ότι τέτοιου είδους όπλα θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε πολύ μακρινές καταστάσεις. Α, παρακαλώ. Α, κύριε Άλλη, συγγνώμη, συγγνώμη, παρασύρθηκα από τα πυρηνικά, βλέπετε, και κόντεψα να ξεχάσω τη δικιά σας την ερώτηση. Ρωτήσατε για τον την νότια πτέρυγα. Ναι, υπάρχει μια διευκόλυνση που την ε, ε, αναπτύσσουμε τώρα. Θα υπάρξει συνάντηση στην Νάπολη και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα για παρετέρω συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε ότι θα είναι μια διευκόλυνση που θα μας επιτρέψει να συγκεντρώσουμε πραγματογνωμοσύνη και σε στρατιωτικά αλλά και σε μη στρατιωτικά ζητήματα οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που έχουν να προτείνουν πραγματογνωμοσύνη από τον ακαδημαϊκό χώρο, για παράδειγμα, επειδή έχουν εμπειρογνώμονες από τη Μέση Ανατολή και μπορούν να μας βοηθήσουν στην ανάλυση μας στην Απόλη είναι ευπρόσδεκτοι. Είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα συνεργασίας, λοιπόν, ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι μια καταπληκτική νέα ικανότητα που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για νέες ε, επιχειρήσεις. Και θα συζητηθεί και στη διάσκεψη σίγουρα. Ευχαριστώ. Η απάντηση του κυρίου Σεράνου τώρα παρακαλώ. Συνήθως είναι συμπληρωματικές οι απαντήσεις σα. Ε, είχατε και αρκετέ ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και φυσικά προσυπογράφω όσα είπε η Ροζ, όσον αφορά την απειλή για τι αξίε μα. Νομίζω ότι επειδή επευθύνεται την ερώτηση ε, σε ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους σε εξωτερικές σχέσεις και στις, ε, ε, σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και νομίζω ότι η απάντηση πρέπει να έρθει από αυτή την οπτική γωνία. Καταρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφώς ποια είναι η εξωτερική διάσταση όλων αυτών ε, τα οποία θεωρούνται ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ξενοφοβία. Να εξηγήσουμε δηλαδή ποιες είναι οι απειλές ε, στο μέτρο του δυνατούν και τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές. Διότι η ξενοφοβία σίγουρα ποτέ δεν θα είναι απάντηση και ε, υπάρχει ευθύνη να διαβιβάσουμε και αυτό είναι το δικό μας το αφήγημα που έχουμε να αντιτάξουμε ε, πρέπει να εξηγήσουμε και να δούμε πώς βλέπουμε εμεί τα πράγματα και τι απάντηση παρέχουμε και ε, η ξενοφοβία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απάντηση στις απειλές ε, που είτε είναι πραγματικές είτε αντιλαμβάνεται ως πραγματικές ο κόσμος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει ε, όσον αφορά την αποτροπή πυρηνικών απειλών, ε, νομίζω ότι αυτό είναι τομέα τη ε, Rose. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με αυτό. Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε στους αντιπάλους ε, τι στόχους έχουμε και τι όρια υπάρχουν, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπεραστούν και νομίζω ότι σαφείς στόχοι και σαφείς προθέσεις ε, πάντα βοηθούν στις διεθνείς σχέσεις. Δεν θα επισέλθω βέβαια στα τεχνικά θέματα, διότι δεν είμαι η δήμον για να απαντήσω, ε, ιδίως όταν είναι ροή στην αίθουσα. Όσον αφορά την νότια πτέρυγα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εκεί υπάρχει δουλειά για όλους, ε, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές προκλήσεις και θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με τον ΝΑΤΟ για να εξηγήσουμε τι κάνουμε εμεί σε κάποια θέατρα επιχειρήσεων και πώ μπορούμε να συνεργαστούμε σε κάποια άλλα θέατρα επιχειρήσεων. Νομίζω ότι η Ρόζα αναφέρθηκε και σε αυτό προηγουμένω. Ο συνδυασμό των μέσων που διαθέτουμε και τι έχουμε να προσφέρουμε θα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι εν τέλει θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο σύνολο δυνάμεων. Και ό,τι και να κάνουμε, ε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι κοινά και θα είναι συνήθως κοινά και για τους δύο οργανισμούς. Επομένως, αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, ε, το πώς θα αντιλαμβάνονται οι χώρες που βοηθούμε τα θέματα αυτά και το γεγονός ότι ό,τι συνδρομή δίνουμε πρέπει να είναι κατόπιν αιτήσεων και, αιτήσεως και να είναι ευπρόσδεκτη. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να του βοηθήσουμε καλύτερα αλλά προσβλέπουμε και στο πώς θα προχωρήσει, πώς μπορούμε να το συνεχίσουμε, πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία. Για τα Δυτικά Βαλκάνια, Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το θεματολόγιο και ενδείξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις έγινε και η Σύνοδος των Δυτικών Βαλκανίων και προσπαθούν να προχωρήσουν το θεματολόγιο αυτό με όλους τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και βεβαίως είναι και πολύ σημαντικό τμήμα της λύσης. Και ο ρόλος του ΝΑΤΟ βεβαίω είναι εξίσου σημαντικός και πολλές από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, έχουν ενταχθεί ή είναι στη διαδικασία ένταξης ε, στο ΝΑΤΟ Μόνο μία βέβαια εντάχθηκε προσφάτως. Αλλά αυτό είναι ένα θεματολόγιο με το οποίο συμφωνούμε και το υποστηρίζουμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον αναφέρεστε σε ε, επιπλέον ε, ε, μέλη δεν έχουμε έξοδο από τον ΝΑΤΟ, δεν περιμένετε κάτι τέτοιο, να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Λεκλουά από το Βέλγιο και μετά τον κύριο Νέβης από την Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γαλλικά. Εξεπλάγει ευχάριστα από την παρέμβαση του κυρίου Σεράνο προηγουμένως, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ευρώπη της Άμυνας και αυτό δεν είχε καμία αντίφαση με τα σχέδια και τις ε, ε, προβλέψεις του ΝΑΤΟ, γιατί φυσικά ορισμένες φορές μπορεί και να αποτύχουμε, γιατί έχετε και το στένος να πείτε ότι ακόμα και αν είμαστε φίλοι και σύμμαχοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν ε, αποκλήσεις και απόψεις οι οποίες μπορεί να μην συγκλίνουν. Και επίσης ε, είπατε και το εξήγησε και η κυρία Γκότερ Μουλέρ ότι υπάρχει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε πολύ η κυβερνοασφάλεια και όσον αφορά τα πλαίσια της συνεργασίας αυτής της διάσκεψης, διάβασα και το έγγραφο το οποίο μας εδόθηκε, το πολύ καλογραμμένο έγγραφο της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, που μας έδωσε η Γραμματεία και εδώ λέει ότι υπάρχει ένα δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 η Μαΐου του 2018 που είναι πρόσφατο δηλαδή που εξηγούσε ότι η δυσκολία που έχουμε σε θέματα κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός σε εθνικό επίπεδο των στρατηγικών και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιαμφισβήτητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να ενισχύσουμε την εσωτερική συνεργασία αλλά και την εξωτερική συνεργασία με το ΝΑΤΟ όπου υπάρχει εκεί τεχνογνωσία ε, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα λοιπόν να σας επισημάνω ε, τι πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Να τονίσω επίσης ότι, ε, και δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά στην Ευρώπη, τουλάχιστον στη χώρα μου, ορισμένες φορές Υπάρχει σπάνιδα αυτής της εξειδίκευση ε, των αναλυτών του κυβερνοχώρου ε, και κυρίως σε εγκληματολογικά ζητήματα και επομένως πρέπει να δούμε και τι δυνατότητες έχουμε να βελτιώσουμε τις συνέργειες διότι πολύ συχνά διαπιστώνω ότι επικεντρωνόμαστε και δεν είμαι και από μια χώρα που είναι και ο καλύτερος μαθητής ε, διότι δεν είμαστε από αυτούς που δίνουμε το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα αλλά ε, ορισμένες φορές υπάρχουν συνέργεια και σε αυτή την περίπτωση και ενίσχυση της συνεργασίας θα μπορούσε να βοηθήσει και να έχει μια ενδιαφέρουσα προστιθέμενη αξία, κυρίως ε, ε, σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται σε αυστηρά όρους προϋπολογισμού, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουν οι χώρες και τα θέματα προϋπολογισμού και σε οικονομικό. Επομένως, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε επιλογές στον προϋπολογισμό. Πώς ε, θεωρείτε εσείς λοιπόν ότι πρέπει να ενισχύσετε την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα κυβερνοεσφάλειας ε, και σε σχέση με το ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς βλέπετε τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αντίστοιχα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τελειώσω και την παρέμβαση διότι ήδη μακρηγόρησα και να ε, ρωτήσω πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη διάθεση που εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές στη συνεδρία στην Επιτροπή τους για την σύσταση αυτής της Ευρωπαϊκής Ομάδας ταχείας αντίδρασης σε θέματα κυβερνοασφάλειας που θα μπορούσε να ε, διαπιστώσει, να ανοιχνεύσει φυσικά την, ε, ε, κάποια κυβερνοεπίθεση. Να συγχαρώ φυσικά και τους ευρωβουλευτές οι οποίοι μετά όσα κάνουν στην Αρμόδια Επιτροπή κατάφεραν να συμφωνήσουν με αυτό που προσπαθούν να πετύχουν οι πελίτες. Επομένως ένα μεγάλο μπράβο από μένα. Ευχαριστώ αλλά να πω και ότι η έκθεση που είδα στην Βαρσοβία για τις νέες τεχνολογίες και την κυβερνοασφάλεια ήταν εξαιρετική, σε εξαιρετικό επίπεδο που είχε ε, συνταχθεί από, ε, από βουλευτές συναδέλφους. Θα δώσω το λόγο για μερικές ακόμα παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και την κυρία Γκότερ Μίλλερ και τον κύριο Πέντρο Σεράνο που είναι εδώ σήμερα και απαντά στις ερωτήσεις μας τρεις ερωτήσεις που έχουν ένα κοινό στοιχείο. Προσπαθούν να διευκρινίσουν διάφορες έννοιες. Πρώτον, ο Αντιπρόεδρος Πάσκου πριν από μία ώρα είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική σημασία και ευρωπαϊκή συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των συνθήκων θα έχει, προσπαθεί να έχει μονάδες μάχης. Ε, υπάρχει μια στρατιωτική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δηλαδή μια στρατηγική αυτονομία που δεν ξέρω ακριβώς ε, περί τίνος πρόκειται. Αν θα μπορούσατε λοιπόν κυρίως ο κύριος Σεράνο να μας διευκρινίσει αυτή την έννοια και ε, την προσέγγισή σας, ε, θα σας ήμουν ευγνώμων. Δεύτερον, για, τη την νότια πτέρυγα. Είναι πολύ εύκολο να λέει κανείς νότια ε, πτέρυγα και νότος, αλλά συνειδητοποίησα ότι ο νότος για διάφορες χώρες σημαίνει κάτι διαφορετικό ο Νότος ε, είναι και μια περιοχή, μια πολύ μεγάλη περιοχή που περιλαμβάνει και τη Βόρεια Αφρική. Αλλά ο Νότος είναι και η περιοχή του Σαχέλ. Και παραπέρα και πιο βαθιά νότια. Και αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι ε, από ό,τι φαίνεται στα νότια της Βόρειας Αφρικής ε, είναι σαν ε, ε, no man's land, σαν να μην κατοικείται από κανέναν, σαν να μην ανήκει σε κανέναν. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται λοιπόν με όλο αυτό το θέμα της ευθύνης προς τους γείτονες και όσον αφορά την αμυντική προοπτική, τη βαθύτερη Αφρική, αν μου επιτρέπετε τη χρήση του όρου. Διότι έχω την εντύπωση ότι ε, τείνουμε να λέμε ότι αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών και όχι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ευθύνη του ΝΑΤΟ. Και η τελευταία ερώτηση είναι η διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ σημαντική έννοια, μεν, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, την οποία δεν διαθέτουμε και μπορεί να υπάρχει μια κάποια διαμάχη μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών και αν πάτε και στην περιοχή του κόλπου θα δείτε ότι υπάρχουν ε, ε, διάφοροι οι οποίοι προσπαθούν να πουλήσουν αμυντικό υλικό σε, στις χώρες αυτές σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις ε, μόνο. Είναι τελευταία σας ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις. Ποιος άλλος λοιπόν θα ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση. Κάποιος που ήρθε αργότερα. Όχι. Εγώ έχω μια ερώτηση. Στην πληρωματική προς τις ε, δικές σας. Θεωρείτε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συμμάχων ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ένταση μεταξύ των συμμάχων αυτών, ε, έχει περιθώρια βελτίωσης, ε, καθώς είναι αναγκαίο να υπάρχει όχι μόνο κυβερνασφάλεια, αλλά και να μειωθούν οι δαπάνες με, στα σύνορα συμμάχων. Ενώ πρέπει να αυξηθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων μας. Κύριε Κιώτα έχετε το λόγο. Πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Κύριε Λακουάμα, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας, παρότι τα γαλλικά μου δεν είναι και τόσο καλά, να σας ευχαριστήσω λοιπόν ε, για τα λόγια σας και την παρέμβασή σας. Η έκθεση για την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ ήταν μια πολύ καλή και ισχυρή έκθεση και νομίζω πως ε, και η Ολομέλεια στο Στασβούργο έδειξε πως ε, έχει γίνει καλή δουλειά και είναι ενδεικτική η έκθεση του τι προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες ερωτήσεις σας, για παράδειγμα την ε, κυβερνοάμυνα και την συνεργασία στον κυβερνοχώρο, αυτοί είναι τομεί στους οποίους δεν σταθήκαμε ούτε εγώ ούτε ο Πέτρο αρκετά προηγουμένως και είναι ένας τομέας ε, όπου υπάρχει πραγματικό δυναμικό για ε, σημαντική και καρποφόρο συνεργασία. Υπάρχει, υπάρχουν διάφορες μορφές ε, βιομηχανικής εταιρικής σχέσης ε, για την κυβερνασφάλεια, οι οποίες αφορούν την έγκαιρη προειδοποίηση ε, για επιθέσεις, για την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο στο σύνολο όσο και στις επιμέρους χώρες συμμάχους του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν και πολλά τεχνικά στοιχεία βέβαια, τεχνικές λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί αυτή η καλή συνεργασία. Όμως ε, γίνονται πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. Και από την οπτική γωνία τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ πως αυτοί είναι τομείς στους οποίους ε, μπορούμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και να επαναλάβω ότι όταν ήμουν στη Σιγκαπούρη, στο Σαγκριλά, στο πάνελ που συμμετείχα, συζητήθηκε η νέα ε, τεχνολο... Ε, τεχνητή νοημοσύνη και οι άλλες καινοτομίες, όπως για παράδειγμα κρυπτογράφηση, ε, quantum computing και όλα αυτά τα οποία θα μας φέρουν πιο μπροστά και θα βοηθήσουν στην παροχή καλύτερης, καλύτερων υπηρεσιών άμυνας, κάτι το οποίο θα ωφελήσει και την κοινωνία μας στο σύνολό της. Υπάρχουν όμως και, άλλα, και άλλες αρνητικές πτυχές της πρόοδου αυτής, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να χαλιναγωγήσουμε αυτήν την πρόοδο και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις προκλήσεις όχι μόνο για τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων αλλά και μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά δεν μπορώ να τονίσω αρκετά τη σημασία που έχει η συνεργασία με τη βιομηχανία μας σε όλη αυτή την εξίσωση. Είναι πολύ σημαντική και θεωρώ πως ε, εδώ υπάρχει πολύ, ε, θετική, πολύ θετικό κλίμα. Τώρα, ε, τα σχόλια του συναδέλφου από την Πορτογαλία. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτά. Ε, κάποια από αυτά προορίστηκαν για τον κύριο Σεράν, οπότε λοιπόν ε, δεν θα τα σχολιάσω, αλλά να πω ότι είναι πράγματι μια πρόκληση ε, το πόση προσοχή δίνουμε στο Νότο. Πάντα το ΝΑΤΟ είχε έμφαση στη Μεσόγειο και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όμως αναγνωρίζουμε ότι αναδύονται απειλές και πιο νότια από αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε την περιοχή του Σαχέλ και τον βαθμό στον οποίο χρειάζεται ε, να δώσει προσοχή το ΝΑΤΟ στα τεκτενόμενα εκεί. Όχι μόνο εκεί, αλλά ακόμα και πιο νότια, στον κόλπο της Γουινέας, όπου παρατηρούμε έντονα φαινόμενα πειρατείας και παρόμοιας ε, οικονομικής δραστηριότητας, μαύρης οικονομικής δραστηριότητας, ε, που δημιουργούν αστάθεια και δημιουργούν όχι μόνο αλλά και προσφυγικές ροές από τις περιοχές αυτές. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς με τους ε, περιορισμούς που έχουμε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, ε, διότι οι προκλήσεις αφορούν όχι μόνο τα διαθέσιμα μέσα, αλλά είναι και γεωγραφικές. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε λίγες αλλά σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας, για παράδειγμα με την Αφρικανική Ένωση, η οποία συνεργάζεται πολύ καλά όχι μόνο με τον ΝΑΤΟ αλλά και ε, με άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς και νομίζω πως υπάρχει ευκαιρία σταδιακά και λέω σταδιακά πάλι δεδομένων ε, των οικονομικών μας πόρων να βελτιώσουμε τη συνεργασία διότι υπάρχουν απειλές που μπορεί να αποβούν πολύ σοβαρές ε, για την ε, Μεσόγειο και την ευρύτερη ε, περιοχή της Ευρώπης που προέρχονται από την Αφρική, από αυτές ακριβώς τις περιοχές. Μετά, η διάδραση και η αμυντική βιομηχανία, αν δεν κάνω λάθος, εκεί σταθήκατε. Να πω πως η διαλειτουργικότητα είναι στο κέντρο της συμμαχίας μας και πως ε, τα μέλη του ΝΑΤΟ κάνουν αγορές από άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να δώσουμε την δέουσα σημασία στη διαλειτουργικότητα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε ε, περισσότερο αποτελεσματικοί στη διασφάλιση της ε, ασφάλειας και της άμυνας. Τώρα, στην άλλη ερώτηση, να πω ένα ξεκάθαρο όχι. Βλέπουμε τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, βλέπουμε το πώς ε, χειρίζονται διάφορες ασήμαντες ε, επικοινωνίες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε, διότι αυτό σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της ε, ίδιας της συμμαχίας μας. Όπως είπα και πριν, βρίσκεται στην καρδιά τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της αμυντικής βιομηχανίας. Είναι απολύτως απαραίτητη η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η περίπτωση όπου εισάγονται συστήματα εκτός ΝΑΤΟ εκτός της αμυντικής βιομηχανίας του ΝΑΤΟ και στην περίπτωση αυτή πρέπει να δούμε προσεκτικά τη διαλειτουργικότητα, διότι υπάρχουν εύλογες ανησυχίες για το την ε, μακροβιότητα της, ε, των ε, προγραμμάτων αυτών και των συστημάτων. Επίσης, η Πρόεδρος ρώτησε για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συμμάχων. Για να είμαι ειλικρινής νομίζω πως ε, ο τομέας στον οποίο πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και θα το σταματήσω εδώ για να δώσω το λόγο στον Πέδρο στα πλαίσια της αύξησης της ε, συνεργασίας μας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμβεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ε, σημαντικές προκλήσεις που υπάρχουν και να βρούμε τρόπο για να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών και μεταξύ συμμάχων, άλλωστε. Αυτό το θεωρώ ως ε, κύρια προτεραιότητα δική μας και φυσικά πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα εάν θέλουμε να υποφεληθούμε από το 100% των ε, προγραμμάτων και των ε, σχεδίων που τρέχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο κύριος Σενάρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λακροά, για την ερώτησή σας. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο κλάδο για μας. Εφόσον τον ονομάσουμε κυβερνοάμυνα. Για την κυβερνοασφάλεια αυτό είναι κάτι με το οποίο έχουμε ασχοληθεί ήδη. Με σημαντική συνεισφορά. Έχουμε την οδηγία της νίκης για παράδειγμα που αποτελεί βασικό στοιχείο για να καθορίσουμε προδιαγραφές που βοηθούν την ασφάλεια των διαφόρων συστημάτων στον κυβερνοχώρο. Τώρα, τα όρια ανάμεσα στην κυβερνοασφάλεια και την κυβερνοάμυνα δεν έχουν οριοθετηθεί ακόμα απόλυτα. Και γνωρίζετε και την κοινή ανακοίνωση, η οποία παρουσιάστηκε πότε, τον Οκτώβριο, αν δεν απατώμε, που μας πέρασε. Παρουσιάζει διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ενδεχομένως σε δομές οι οποίες με τη σειρά τους να καταλήξουν σε δομές κυβερνόμενας. Προς το παρόν πάντως υπάρχει η ασφάλεια των θεσμών, των θεσμικών οργάνων που είναι ήδη μια δυσκολία, η προστασία των αποστολών μας, των αντιπροσωπιών μας, των εγκαταστάσεών μας εδώ στις Βρυξέλλες ή αλλού. Οπότε όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο σημαντικών προσπαθειών για να ενισχυθεί η ασφαλειά τους ακριβώς. Και μετά είναι και τα κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε σε μια πρωτοβουλία στα πλαίσια της δομημένης συνεχισμένης συνεργασίας που προβλέπει τη δημιουργία ομάδων που θα μπορούσαν να παρέμβουν σε περίπτωση κρίσης. Άρα υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που προχωράνε. Φιλόδοξα προγράμματα επίσης ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο. Τώρα είμαστε στο στάδιο της ε, τελικής ε, διαμόρφωσης. Για το κατά πόσο τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στρατιωτικό σύμμαχος, οπότε τι κάνει με την άμυνα και την ασφάλεια, θα προσπαθήσω να αρχίσω από τον Νότο, που αποτελεί ένα παράδειγμα του τι κάνει επιχειρησιακά. Γιατί ο Νότος δεν είναι no man's land, είναι ένας χώρος όπου δραστηριοτείται όλος ιδιαιτέρως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια. Και θα έρθω σε κάτι που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε σαν ζώνη ασφάλειας, έτσι, από τη Σομαλία, ε, όλο το Σαχέλ. Οπότε εδώ, ναι, πρόκειται για δράσεις ασφάλειας με διάφορα μέσα στήριξη κυβερνήσεων, ανάπτυξης, αλλά και δομές ασφάλειας και στήριξη προσπαθειών που κάνουν οι Αφρικανοί εταίροι μας. Το έκανε το G5 Σαχάρα, στη Σομαλία, με το Σόφια, άλλες προσπάθειες που κάνουμε από κοινού με τον ΟΙΕ, στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, πολλές προσπάθειες και οικονομικές αλλά και ανάπτυξης αποστολών εκεί. Έχουμε πάνω από 500 στρατιωτικούς στο Μαλί που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα για να βοηθήσουν τις επιτόπου δυνάμεις στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ανάμεσα στο Μαλί και τον Νίγηρα Έχουμε 200 αστυνομικού που στηρίζουν τι αντίστοιχε δυνάμει των χωρών αυτών. Έχουμε κάπου 150 στρατιωτικού επίση στη Σομαλία. 60-70 αστυνομικού. Έχουμε και στις ακτέ, ναυτική δύναμη της Σομαλίας και για να αντιμετωπιστεί η πειρατεία αλλά και για γενικότερους λόγους ασφάλειας. Έχουμε Επίσης στήριξη στη Λιβύη που αποτελεί στοιχείο κλειδί όπως ξέρετε ε, του συνόλου της Σαχέλ επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ασφάλεια και άρα επιδρά αρνητικά ε, στις χώρες Σαχέλ. Έπειτα η παράνομη διακίνηση πηγαίνει από το Σαχέλ στη Λιβύη και φτάνει στην Ευρώπη. Συνεπώς, έχουμε αναπτύξει μία μη στρατιωτική αποστολή Βέβαια τώρα για τη Λιβύη ολόκληρη συζήτηση θα μπορούσε να κάνει κανείς. Πάντως εμείς αυτό το κάναμε για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση εθνικής Εθνική Συμφωνία στην Λιβύη με στοιχεία νοικοδόμησης, ασφάλειας και έχουμε και ένα αυτιλιακή αποστολή στην Κεντρική Μεσόγειο η οποία αναπτύχθηκε για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα την ε, μεταφορά, την εκμετάλλευση και μεταφορά ε, μεταναστών και προσπαθούμε επίσης και για την επιβολή του εμπάργου όπλων αλλά και για να αποφύγουμε το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Πολλές λοιπόν από τις προσπάθειες που έχουν αναπτυχθεί επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτά που λέτε. Και γι' αυτό σας περίγραψα και για τον Νότο, έτσι, και η Κεντρική Αφρική εκεί έχουμε στρατιωτική εκπαιδευτική δύναμη για το στρατό εκεί. Λοιπόν, πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε επικεντρώνονται στον Νότο. Θα παρουσιάσουμε και πιο φιλόδοξες προτάσεις στο μέλλον για να στηρίξουμε τις χώρες Σαχέλ G5, να στηρίξουμε την κοινή τους δύναμη, αυτή που δημιούργησαν δηλαδή, αλλά και σε εθνικό επίπεδο για να ενισχύσουν τις δικές τους ικανότητες ασφάλειας και ναυτιλιακά. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Τώρα, δείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και την άμυνα. Μπορούμε να το συνοψίσουμε σε πέντε στοιχεία. Οι ικανότητες άμυνας, ανάπτυξη δηλαδή αμυντικών ικανοτήτων. Ανάπτυξη ε, δομών για την αντιμετώπιση κρίσεων δικών μας. Είναι αμυντική πολιτική αυτή αυτή. Αντιτρομοκρατία, κυβερνοάμυνα, ε, στη θάλασσα, ε, άμυνα και συνεργασία με τους εταίρους μας. ΝΑΤΟ σίγουρα, κυρίως με το Ηνωμένο Έθνη είναι κύρια εταίρεια, αλλά και διμερός με άλλους εταίρους. Και το άλλο είναι επιχειρήσει και στήριξη σε διάφορες χώρες. Ναι, κάνουμε πράγματα στην ασφάλεια για την άμυνα, αλλά τα κάνουμε σε συνδυασμό με την προσέγγιση της κάθε χώρα. Γι' αυτό μιλάμε και για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε χώρε στο Σαχέλ. Τι σημαίνει αυτό. Δεν τους βοηθάμε μόνο την ασφάλεια και την άμυνά τους, τους βοηθάμε και για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια, μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το εμπόριο. Πρόκειται δηλαδή για ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων ε, στήριξης προς αποτροπή συγκρούσεων και προκειμένου οι χώρες αυτές να είναι λιγότερο ευάλωτες και έφραστες. Αυτά κάνουμε λοιπόν για την ασφάλεια και την άμυνα συνεργασία με την Αφρικανική Ενότητα. Βεβαίως. Μόλις υπογράψαμε ένα νέο μνημόνιο κατανόητησης για συνεργασία μαζί τους. Έχουμε διαβουλεύσεις δύο φορές το χρόνο σε επίπεδο πρωτευουσών για θέματα κλειδί. Για τις άλλες ερωτήσεις λίγα έχω να προσθέσω σε αυτά που τα σημαντικά που ήδη είπε για να πληρωτήσει Γενική Γραμματέας για το Μελερ για την ε, διαλειτουργικότητα. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι αμυντικές ικανότητες πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επαφή, επικοινωνία και διάδραση με τις άλλες χώρες. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις και στη Μεσόγειο, διότι είναι και σταυροδρόμοι. Και ο Παόλο Άλλη έχει και την εξής πρόκληση ως Ιταλός με τη Λιβύη. Επομένως αυτή θα είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν οι ομιλωτές, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εκτιμούμε για την παρουσία τους και για το γεγονό ότι απάντησαν σε όλε τι ερωτήσει. Δεν απέφυγαν ούτε μία, ήσασταν πολύ τολμηροί και ειλικρινοί στι απαντήσει σα και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ε, ε, είναι πάντα το αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν ε, ε, δεν έχετε κάποια άλλη υποχρέωση, πολύ θα ήθελα να βρεθείτε και στο επόμενο πάνελ. Θα κλείσει ο Πάολο αυτό το πάνελ και θα κάνει την εισαγωγή το επόμενο. Δεν ξέρω αν θα μείνετε μαζί μας. Εντάξει, καταλαβαίνω. Απαντήσετε σε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Uh, Great meeting.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με το δεύτερο πάνελ του σεμιναρίου. Μετά τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ε, με τον κύριο Σεράνο και την κυρία Γκότεν ε, θα ήθελα τώρα να περάσουμε στον επόμενο μιλητή μας, τον αντιστράτηγο Γιάνν Μπρούξ, ο οποίος είναι αναπληρωτής, ε, ε, είναι γενικός διευθυντής συγγνώμη, του ε, Διεθνού Στρατιωτικού Επιτελείου του ΝΑΤΟ. Είναι Ολλανδός στρατηγός με αξιομνημόνευτη στρατιωτική καριέρα και ως επικεφαλής του επιτελείου είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις μεταξύ των ηθινόντων της σημασίας του ΝΑΤΟ, των δύο στρατηγικών διοικητών, σχέσεις με χώρες εταίρου που εργάζονται στην Ευρώπη και ε, το ε, επιτελείο το οποίο στηρίζει τον Γενικό Γραμματέα και το Διατλαντικό Συμβουλίο για το ε, να προσφέρει την καλύτερη δυνατή συμβουλές πολιτικές, πολιτικής σε θέματα αυτά. Ο στρατηγός Μπρούξ θα παρουσιάσει την εφαρμογή των νέων καθηκόντων που απορρέουν από τις νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας. Δέχτηκε να παραμείνει για ερωτήσεις μετά από την παρουσίαση του. Στρατηγέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ευγενική εισαγωγή. Ε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι ε, εκπρόσωποι, καλησπέρα σας. Ε, είναι τιμή για μένα να ανταλλάζω απόψεις για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσω από τις πιο γενικές παρατηρήσεις που έκανε η αναπληρωτής Γενική Γραμματέας προηγουμένως, αλλά επίσης θα σταθώ όπως ε, τονίστηκε και περισσότερο ε, σε θέματα στρατιωτικής κινητικότητας και φυσικά όπως ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος είμαι διαθέσιμος ε, για ερωτήσεις για θέματα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ αρκεί να παραμείνω στο στρατιωτικό κλάδο γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητά μου. Είμαι πολύ ικανοποιημένο ως Γενικός ε, Διευθυντής ε, από τη θέση στην οποία βρίσκομαι και ε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν άφθονες δυνατότητες να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε περαιτέρω τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις επίσημες σχέσεις σε στρατιωτικό επίπεδο, μας δεσμεύουν συγκεκριμένες συμφωνίες και υφιστάμενες ε, συμφωνίε ε, σε θέματα ασφαλεία. Όσον αφορά το δικό μου το επιτελείο, το Διεθνέ Επιτελείο του ΝΑΤΟ ε, και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε περισσότερο περιθώριο ευελιξία. Όσον αφορά το στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα συναντήσετε αύριο και το Γενικό Διευθυντή και εγώ θα έχουμε πολύ σημαντικές επαφές. Γίνονται ανταλλαγές στη διάσκεψη των Γενικών Διευθυντών και εκεί υπάρχει συμμετοχή όλων των διευθυντών από τα αντίστοιχα επιτελεία και ε, των αξιωματικών από το επιτελείο μας. Είμαι πολύ ικανοποιημένο λοιπόν με τις επαφές ε, μεταξύ επιτελείων ε, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας είπα και προηγουμένως, θα ήθελα να σταθώ σε θέματα στρατιωτικής κινητικότητας περισσότερο είναι ένας από τους βασικούς τομείς τους οποίους ε, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητούν συνεργασία και εδώ θα πρέπει να πω ότι πρέπει και να συνεργαστούμε από αυτόν και θα θυμάστε ότι το ανέφερε και ε, ο Γενικός Γραμματέας ε, στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ πριν από μερικές μέρες στη Βαρσοβία. Από πλευρά μου υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε για τις απαιτήσει, τα πρότυπα και την ε, ετοιμότητα και την ταχύτητα στην ε, κινητοποίησή μας. Οι συγκεκριμένε απαιτήσει, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, μεταφορά των υποδομών, είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, το λογικό είναι να είναι κοινά και την έχω ξανακούσει αυτή τη φράση, να έχουμε ένα κοινό σύνολο δυνάμεων. Και επομένως, κατά την άποψή μου, είναι υψή της σημασίας και οι δύο οργανισμοί να συμφωνήσουν, να ευθυγραμμίσουν τις ε, σχετικές στρατιωτικέ απαιτήσει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα κοινό σύνολο απαιτήσεων. Ε, από αυτή την άποψη, οι επικεφαλής ε, της άμυνας συναντήθηκαν στην Στρατιωτική Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ αργότερα και αναγνώρισαν την πρόοδο που έγινε μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, αναφέροντα και το ε, πώς συμβάλλει το ΝΑΤΟ όσον αφορά τι στρατιωτικέ απαιτήσει στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, υπήρχε η συμβολή του ΝΑΤΟ όσον αφορά τι στρατιωτικέ απαιτήσει στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, στρατιωτική κινητικότητα. Ε, κυρίως ζητάμε περαιτέρω στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης ε, ε, να συμπεριληφθούν και μη Ευρωπαίοι σύμμαχοι στη διαδικασία ευθύς εξ αρχής. Οι επικεφαλεί τη άμυνα τόνισαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διαδικασία συντονισμού προκειμένου να εξασφαλίσουμε και συνοχή στι απαιτήσει και να συνεχίσουμε να το εξασφαλίζουμε αυτό στη συνέχεια. Μπορώ να σας πω ότι στη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς ε, το στρατηγείο του ΝΑΤΟ σε επίπεδο επιτελείου κατάφερε να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ε, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνας ε, στη συνεργασία για τη διασυνοριακή κινητικότητα και μεταφορά και πιο πρόσφατα το επιτελείο μου συναντήθηκε με το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά μια κοινή πρόταση για τις στρατιωτικές απαιτήσει. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι τα πρότυπα για ε, να είναι αποτελεσματικές οι στρατιωτικές απαιτήσει, πρέπει να υπάρχουν πρότυπα και αναφερθήκατε στη διαλειτουργικότητα φυσικά στο προηγούμενο πάνελ. Θα ήθελα εδώ να πω ότι η χρήση των ευρωπαϊκών ε, προτύπων για να καθορίσουν τις απαιτήσεις ε, χρησιμοποιούν ε, μια αποτελεσματική, συμφωνημένη, καλά χαρτογραφημένη διαδικασία και ένα σύστημα το οποίο έχουν επαληθεύσει και πάρα πολλές χώρες εταίρει. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι τα πρότυπα του ΝΑΤΟ μπορούν να ε, προσφέρουν μια τάξη στη στρατιωτική κινητικότητα και εγώ τι έκανα, έδωσα όλα τα ε, πρότυπα που εφαρμόζουμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ στο επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, ταχύτητα στην κινητικότητά μας. Και εδώ δεν αφαιρόμαστε στο πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί ένα φορτηγό όχημα ή πόσο γρήγορα μπορούμε να περάσουμε φραγμούς, αλλά ε, κυρίως τις αρχές και την ομοθεσία. Το ΝΑΤΟ ασχολείται με το θέμα αυτό, ε, είναι μακροχρόνιο και το 2015 οι σύμμαχοι συμφώνησαν να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες τους, ώστε να επιτρέπεται η ταχεία κινητοποίηση ε, των κοινών δυνάμεων και την ενισχυμένη ε, ειρηνευτική δύναμη σε καιρό ειρήνης. Είναι θετικό αυτό το βήμα, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες από το επίπεδο της λάψης αποφάσεων ε, στις εθνικές ε, κυβερνήσεις μέχρι τον ε, φύλακα στα σύνορα. Είναι πολύ μεγάλη η πορεία και πρέπει κάπως να γίνουμε καλύτεροι και να γίνονται αυτά πιο γρήγορα. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να αναρωτηθούμε πώς οι ικανότητες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμβαδίσουν ώστε να βελτιώσουμε τη δυνατότητά μας να ενισχύσουμε τα πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρέπει να δούμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για τη μηβαία και τη ρήτρα αμοιβαία ε, συνδρομή και αλληλεγγύη τη Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώ μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το άλλο. Απ' τη μια, το άρθρο 222 της Συνθήκης Λειτουργίας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει να ζητηθεί η βοήθεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Από την άλλη, το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε ίσως να δώσει και ένα όχημα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν σε κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης. Η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως δεν είναι ζωτική σημασία μόνο σε περίοδο κρίσης, αλλά εγώ θα μπορούσα να πω και σε περίοδο ειρήνης. Ε, ίσως δε και πιο συγκεκριμένα σε κέντριο γιατί εκεί έχουμε εκπαίδευση, ασκήσεις και γενικότερα ετοιμότητα. Ε, το πιο δύσκολο ίσως σενάριο θα ήταν όταν υπάρχει απέτηση για γρήγορη κινητοποίηση στρατευμάτων, όταν δεν υπάρχουν περιπτώσεις κρίσης ή σύραξης, αλλά θέλουν να αποτρέψουν την κρίση ή τη σύραξη. Ε, για παράδειγμα, η Task Force ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δύναμη ανταπόκρισης του ΝΑΤΟ ε, σημαίνει ότι μπορούμε να κινηθούμε σε περίπτωση κρίσης ή σε περίπτωση άρθρου 5, αλλά οι ανταγωνιστές μας γνωρίζουν ότι ε, υπάρχει αυτό και επομένω προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ταυτόχρονα. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε και εμείς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες μας και σε καιρό ειρήνης, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευέλικτη και ταχεία διαδικασία διαχείρισης και σε καιρό Ελπίζω αυτά τα τρία να σας ε, έδωσαν κάποια στοιχεία για τη συζήτηση, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, είμαι διατεθειμένο να συζητήσω και άλλα στοιχεία της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, Στρατηγέ Πρόξ, για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Δείξατε πολύ σημαντικά θέματα, πιστεύω. Η ταχύτητα της ανταπόκρισης και η κινητικότητα είναι το παν στη σημερινή εποχή και σε έναν κόσμο όπου η ταχύτητα είναι κυρίαρχη. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν για τη συζήτηση και θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μπόσμαν από τις κάτω χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ στρατηγία, ευχαριστώ πολύ για ε, την υπηρεσία σας αυτό τον καιρό. Το ΝΑΤΟ έχει και διάφορα πρότυπα. Όσο υπάρχει το ΝΑΤΟ υπάρχουν και αυτά. Και στόχος είναι να ε, αυξηθεί αυτή η ταχύτητα κινητοποίησης και αυτό είναι και κοινό στόχος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν γίνεται λόγος για τη συνεργασία αρχίζει και υπάρχει ένας εκνευρισμός, διότι λέμε πολλά και δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Τι έχετε να πείτε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να συγκεντρώσουμε πρώτα δύο-τρεις και μετά να προχωρήσουμε στις απαντήσεις. Ωραία. Μπορείτε να απαντήσετε απευθείας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Νομίζω πως ε, θίξατε ακριβώς ε, το σημαντικότερο θέμα. Κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου υπήρχαν κάποια πρότυπα τα οποία εφάρμοζαν ε, όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Υπήρχε οδικό δίκτυο, έτοιμο, ε, λιμένες, ε, αερολιμένες. Ήταν όλα σε τιμότητα. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου όμως χάθηκε αυτό το επίπεδο, αυτή η απέτηση για να υπάρχει το συγκεκριμένο επίπεδο τιμότητας από τα μέλη του ΝΑΤΟ ε, σε στρατόπεδα, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ. Επεκτάθηκε, λοιπόν, επεκτάθηκαν λοιπόν οι επιχειρήσεις μας και ε, ανατολικά. Αυτό ήταν μια εξέλιξη ε, που αφορά τα πρότυπα. Χρειάζεται λοιπόν να τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας σε ό,τι αφορά τα πρότυπα αυτά. Μετά, οι απαιτήσει. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετική αφετηρία όσον αφορά τις απαιτήσει αυτές. Αν ε, δείτε τι προσπαθεί να κάνει το ΝΑΤΟ, θα συνειδητοποιήσετε ότι προσπαθούμε να μετακινήσουμε ε, βαριά οπλισμένη στρατό στην Ευρώπη και πρέπει να φροντίσουμε να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάμεσα στα διάφορα κέντρα. Μετά υπάρχουν και οι μικρότερες μονάδες ε, ελαφρύτερου οπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, αυτό που κάναμε, και θέλω εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα ενός τεθροκισμένου ε, του πεζικού το οποίο μπορεί να είναι δύο φορές ε, βαρύτερο ε, σαν όχημα. Πήραμε λοιπόν αυτό ως ε, δεδομένο και το χρησιμοποιήσαμε στην κατασκευή μιας γέφυρας, για παράδειγμα. Υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το βάρος που μπορεί να, να σηκώσει μια γέφυρα. Κοιτάξαμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή τους κανονισμούς ασφάλειας των μεταφορών. Δηλαδή, μπορείς να μετακινήσεις προσωπικό μέσα σε οχήματα από το σημείο Α στο σημείο Β και ταυτόχρονα στο ίδιο όχημα να μεταφέρονται και ε, πυρομαχικά. Μετά ε, μπορούμε να μεταφέρουμε διαφορετικούς τύπους πυρομαχικών στο ίδιο όχημα. Κοιτάξαμε λοιπόν ε, με μεγάλη προσοχή τους διαφορούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε, διότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να μετακινηθεί ένοπλο προσωπικό μαζί με πυρομαχικά και οχήματα. Εάν θέλεις να μετακινήσεις μία μονάδα εννέα ε, πεζικάριων με τα οχήματά τους, με τον οπλισμό τους, ε, αυτό θα χρειαστεί 24 ώρες. Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος είναι να ε, μετακινηθεί τμηματικά. Αυτό όμως επειδή δεν γίνεται χρειάζεται να βρεθεί μια λύση. Και ε, πρέπει στη λύση αυτή να είμαστε ρεαλιστές. Σίγουρα πρέπει να γίνουν ε, πολλά, πολλές βελτιώσεις. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ και τα θεσμικά όργανα προσπαθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ο πρόεδρος Τούσκ το είπε ότι ε, προσπέπουμε στην επόμενη σύνοδο έτσι ώστε να κληθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να λάβουν αυτές τις ε, υπαρκτές ανησυχίες σοβαρά υπόψη. Μετά, ικανότητα ανταπόκρισης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μπορούμε να στείλουμε μονάδες ε, πολύ γρήγορα, όμως υπάρχουν άλλα προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τώρα, ο συνάδελφος από την Τουρκία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Από όσο γνωρίζω, το Διεθνές ε, Στρατιωτικό Προσωπικό μπορεί να δραστηριοποιηθεί από την ε, αρμόδια, επιτροπή, την αρμόδια αρχή του ΝΑΤΟ. Εσείς είσαστε υπεύθυνο για αξιολόγηση και μελέτες όσον αφορά στρατιωτικά ζητήματα του ΝΑΤΟ που εντοπίζουν στρατηγικά ενδιαφέροντα και προτείνουν και τρόπους δράσης. Στο στάδιο αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τις ρωσικές ε, ικανότητες στην Μεσόγειο. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι οι ρωσικές ε, ικανότητες, όχι στη Μεσόγειο, συγγνώμη, στην Αυτιλία, μπορούν ε, ίσως να επεκταθούν σε θέματα πολιτικής και στρατηγικής διαφοροποίησης. Έτσι το στρατηγικό πλαίσιο γίνεται πιο περίπλοκο και πιο δύσκολο για αυτούς που σχεδιάζουν, πολιτική, αποφασίζουν. Οπότε γι' αυτό θέλω να ρωτήσω ότι έχετε να πείτε για τις ρωσικές ικανότητες ε, στη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εύκολη ερώτηση, λέει αστευόμενος ο μιλητής. Εδώ είναι που πρέπει να κοιτάξουμε συνολικά το θέμα και συγχρόνως τους τέσσερις τομείς που είναι η Μεσόγειος, ο Ατλαντικός, η Βαλτική. Πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα πώς αναπτύσσεται στη θάλασσα η Ρωσία. Υπάρχουν δύο προτεραιότητες. Είναι τα πυρηνικά και είναι η στρατηγική ε, ναυτική ανάπτυξη. Υπάρχει προτεραιότητα όσον αφορά δηλαδή τα κονδύλια, τον προπολογισμό και βλέπετε πώς ε, προχωρούν προς το μέλλον, κυρίως με τα υποβρύχια. τα ξέρετε κι εσείς από την Μαύρη Θάλασσα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ανταγωνισμός στη θάλασσα. Επειδή όταν μιλάμε για τις εξελίξεις στους διάφορους τομείς, μέχρι τώρα στη Μαύρη Θάλασσα ή στη Βαλτική Θάλασσα έχουμε δει παρουσία, έχουμε δει πολλούς πειραματισμούς, ασκήσεις αλλά αυτά που συμβαίνουν στη Βαλτική δεν υπερβαίνουν τις προδιαγραφές που θα περιμέναμε. Στη Μαύρη Θάλασσα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το θαλάσσιο αποτύπωμα εκεί υπερβαίνει αυτό που θα έπρεπε για να ελέγχεται η Μαύρη Θάλασσα. Οπότε βλέπουμε προσπάθεια επιρροής στη Μεσόγειο. Βλέπουμε επίσης στοιχεία όσον αφορά την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Πάλι για την επιρροή, έτσι. Οπότε ναι, χρησιμοποιείται για επιρροή Μαύρη Θάλασσα. Καλύπτω έτσι εν μέρη και τη Μεσόγειο. Ε. Στη Μεσόγειο τους βλέπουμε να κινούνται όλο και περισσότερο, να έχουν παρουσία μερικές φορές βλέπουμε ότι είναι μια δύναμη που θέλει και να καυχηθεί, να μας ε, δείξει ότι προχωράει σε επιρροή εκεί. Προς το παρόν, ε, με τις τωρινές μονάδες χρειαζόμαστε ενίσχυση. Και από την Χερσόνησο προσπαθούμε να επηρεάσουμε την επικοινωνία, γιατί όντως πρόκειται για απειλή για μας. Συνολικά δηλαδή, θα έλεγα, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το τι κάνουν. Και ο κύριο Μίλλερ νομίζω ότι το κάλυψε αυτό. Θα δείτε στην επόμενη διάσκεψη, η κυρία Γκέντε Μίλλερ το κάλυψε αυτό, θα δείτε ότι στην ε, επόμενη διάσκεψη θα συζητηθεί το ζήτημα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου ε, είναι συνέχεια των όσων λέμε τώρα για την ε, θάλασσα. Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίρρηση από την Ρωσία για την ΠΕΣΚΟ, την ε, συνεργασία, την αμυντική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ένα από τα θέματα που θέτει είναι εποπτεία λιμένων και θάλασσας. Εγώ είμαι από την Λετωνία, αναφέρθηκαν πολλά. Μιλάμε και για περισσότερη προσοχή που θα, θέλε, θα έπρεπε να δώσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή μας, στη θάλασσα. Δεν ξέρω λοιπόν η ΠΕΣΚΟ τα κοιτάει αυτά. Είναι δηλαδή ένας άλλος τομέας ενδυνάμεις συνεργασίας. Η ασφάλεια στη θάλασσα το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να ασχοληθεί με την ασφάλεια δηλαδή στη θάλασσα στην περιοχή μας για να ξέρει τι γίνεται εκεί. Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι ελάχιστα γνωρίζουμε τα σχέδια ΠΕΣΚΟ. Μερικά από αυτά προχωρούν από κάποιες χώρες, από ομάδες χωρών. Κάποια άλλα βρίσκονται σε πολύ προκαταρτικό στάδιο. Έτσι όμως όπως το περιγράφεται, εγώ θα έλεγα ότι είμαι υπέρ, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ. Αυτό που θα δούμε είναι από τα κύρια στοιχεία της νέας στρατηγικής για τη θάλασσα του ΝΑΤΟ είναι ότι θα πιέσουμε για περισσότερη ευελιξία στην προσέγγιση. Τώρα έχουμε τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που είναι πιο σταθερά στοιχεία. Θα περιοριστούμε σε έναν πιο μικρό ο οποίος θα αντιδρά βάσει στοιχείων ad hoc. Όταν κυκλοφορούν στη θάλασσα θα βλέπουν τι γίνεται όταν είσαι στον Ατλαντικό, μπορείς να ασχοληθεί και να συνεργαστείς με μεγάλα σκάφη, όταν είσαι αλλού με πιο μικρά. Θέλουμε δηλαδή περισσότερη ευελιξία. Κάτι που ταιριάζει απόλυτα με την ΠΕΣΚΟ, αλλά σας είπα ότι δεν ξέρουμε αρκετά πράγματα για τα προγράμματα ΠΕΣΚΟ προς το παρόν. Παρακαλώ. Στρατηγέ. Έρχομαι από τη Σουηδία, η οποία είναι, έχει δεσμευτεί με την αλληλεγγύη στις συνθήκες. Μπορείτε να πείτε περισσότερα πράγματα για το τι βλέπετε ότι θα μπορούσε να κάνει μια χώρα εταίρος. Για το δικό σας πλαίσιο βέβαια. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά βέβαια, αλλά χωρί να μπω σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολλά θα μπορούσε να κάνει κανεί. Γιατί ξέρετε, με τη Σουηδία και τη Φιλανδία προετοιμάζουμε τα σχέδιά μας για τις επιχειρήσεις μας. Πού βασιζόμαστε για τον προγραμματισμό αυτό. Το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να μπορεί από μόνο του να προχωρήσει σε αυτές τις επιχειρήσεις που αποφασίζει, γιατί αποφασίζουμε αυτόνομα το ΝΑΤΟ και μετά η Σουηδία και η Φιλανδία είναι άλλες χώρες που παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Εφόσον όμως επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν δυνάμεις στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά επιπλέον από αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Και έχουμε, το έχουμε δοκιμάσει αυτό σε πολλές ασκήσεις. Υπάρχει βέβαια και η στήριξη δυνάμεων από διάφορες χώρες. Και μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και δεν είναι μόνο στη θάλασσα. Είναι η άρνηση συμμετοχή στις ασκήσεις, κάτι το οποίο βέβαια μας δυσκολεύει στη Βαλτική. Μπορούμε βέβαια να πάμε από γη στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Οπότε ναι, στήριξη με δυνάμεις, με γη, με συνδυτοποίηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη. Τακτικά. Και ο τρόπος διάδρασης μεταξύ Σουηδίας και Φιλανδίας, μια νέα εξέλιξη δηλαδή που θα συμφωνηθεί αυτή τη βδομάδα σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, θα μας δώσει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τα επιχειρησιακά μας ε, σχέδια με τα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Πολλά γίνονται λοιπόν, γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί κάτι στη Βαλτική θάλασσα χωρίς τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Πολλά γίνονται λοιπόν προς το παρόν. Και βλέπω ότι οι χώρες έχουν δεχτεί νομοθεσία για στήριξη ε, δυνάμεων που περνάνε μέσα από τις χώρες τους. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιες, κάποιον άλλο να Παρακαλώ. Αν δεν έχει κάνει άλλη ερώτηση, έχω ερώτηση εγώ. είναι ενδιαφέρον να μας λέτε εσείς πράγματα ως στρατηγός και να έχετε και φίλους από την Ορβηγία να μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο για να βοηθήσουν τους Ολλανδούς ή τους Ολλανδούς να πηγαίνουν ε, ε, στην Αλβανία για να βοηθήσουν ε, τους τεχνικούς εκεί. Μια ερώτηση περισσότερο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά, παρά στο στρατηγό. Βλέπουμε ότι οι αμυντικές βιομηχανίε μας είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και δεν υπάρχουν πάντα ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και προσπαθούν να έχουν κάτι μοναδικό, εξειδικευμένο, να είναι βέβαιο ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δική τους βιομηχανία θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί απειλή ή παρέχει περισσότερες δυνατότητες. Η προσέγγιση δική μας είναι ότι ξεκινάμε από την προοπτική της διαλειτουργικότητας. Για μας ε, στο στρατό η διαλειτουργικότητα έχει αρκετές πτυχές και θα έρθω και στην αμυντική βιομηχανία. Καταρχάς είναι θέμα νοοτροπίας η διαλειτουργικότητα. Γι' αυτό ε, δημιουργήθηκε αυτή η συμμαχία. Γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρχει η ίδια στάση, η ίδια νοοτροπία. Μετά υπάρχει το δόγμα. Το δόγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να συνεργαστεί ε, ακόμα και αν δεν είσαι συνδεδεμένος, αν δεν υπάρχει τεχνική διαλειτουργικότητα, ε, μπορείς να συνεργαστείς αν υπάρχει το ίδιο δόγμα. Και φυσικά μπορείς να επιτύχεις τα πάντα αν υπάρχει και η τεχνική διαλειτουργικότητα ή κατ' ουσία, όπως είπατε, να υπάρχουν ακριβώς τα ίδια πρότυπα και ο ίδιος εξοπλισμός. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι ιδίω όσον αφορά τον ίδιο εξοπλισμό θα ήταν αδύνατον. Υπάρχει εθνική βιομηχανική πολιτική που υφέρπει, δεν θα το θίξω αυτό, αλλά η δική μας ευθύνη ως στρατός είναι να έχουμε τις κατάλληλες απαιτήσεις. Και και εμείς κάποιες φορές ε, προσπαθούμε να έχουμε λύσεις ε, με ε, περισσότερη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Ε, και φυσικά αν έχουμε τέτοια πράγματα θα έχουμε κάτι παραπάνω όταν είναι κάποιος Ολλανδός ή από άλλη χώρα. Έχουμε δηλαδή ο καθένας κάτι επιπλέον. Προσπαθούμε να τα έχουμε όσο το δυνατό πιο απλά και να μην έχουμε τέτοιες λύσεις που είναι πιο αυστηρές σε εθνικό επίπεδο, διότι μόνο έτσι μπορούμε να διασχίσουμε διάφορες χώρες και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε. Νομίζω ότι το NH90 είναι αρκετή απόδειξη. Έχουμε τελείως διαφορετικούς τύπους από το NH90 από ό,τι χώρες. Δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος φυσικά να δαπανούμε τα χρήματα των φορολογουμένων αυτός. Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα. Είναι σαφές τώρα ότι αυτό είναι απαραίτητο για όλους Απ' τη μια αυτό είναι θέμα κανόνων, δηλαδή είναι νομοθετικό ζήτημα και εδώ είμαστε νομοθέτες, επομένως είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου. Αλλά βεβαίως υπάρχει και αντίκτυπος και στις υποδομές, όπως είπατε προηγουμένως. Και το κόστος των υποδομών, οι νέων υποδομών, ή εξυγχρονισμός ε, υφιστάμενων υποδομών, δεν είναι το ίδιο για κάθε χώρα στην Ευρώπη ή κάθε χώρα του ΝΑΤΟ. Έχει κάνει κάποια εκτίμηση το ΝΑΤΟ για το πόσα χρήματα απαιτούνται, τουλάχιστον σε χονδρικό και γραμμές, για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών υποδομών, ώστε να έχουμε πλήρη κινητικότητα. Και αν ναι, πώς θα πρέπει να γίνει και κατανομή των βαρών ε, στο κόστος αυτός. Διότι ως νομοθέτες νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε επενδύσεις σε υποδομές, αναφερόμαστε σε δισεκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, εύκολα φτάνουμε σε τέτοια ποσά. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαχειριστούμε το διαφορικό αντίκτυπο σε χώρες μέλη και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μπορούσε να υπάρξει κάποια στήριξη και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το εξετάσατε αυτό το στοιχείο, διότι έγινε αυτή η συζήτηση στη χώρα μου με κάποιον και ο οποίος μου είπε ότι εάν στηρίζει την ιδέα της στρατιωτική κινητικότητας, τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να μοιραζόμαστε ε, τα βάρη με άλλες χώρες ε, όταν δεν ενδιαφερόμαστε εμεί για τις υποδομές αυτές. Είναι λεπτό λοιπόν το ζήτημα. Και έχω και μία ακόμα ερώτηση. επιτρέψτε μου λίγο να σχολιάσω αυτό ακριβώς το σημείο, να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο δόθηκε από κάποιους Αμερικανούς ε, σε μια συνεδρίαση που είχαμε. Αυτοί πιστεύουν ότι στη διάρκεια κάποιων ασκήσεων, το να έρθουν οι δυνάμεις τους στην Ευρώπη σημαίνει ότι ο στρατός τους ουσιαστικά χρηματοδοτεί κάποιες ευρωπαϊκές υποδομές και είπαν ότι δεν τους πειράζει να δαπανούν χρήματα για στρατιωτικό επιτελείο, αλλά πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χτίζει τις ευρωπαϊκές υποδομές. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, είναι μεγάλο ζήτημα ή το βγάζουμε εκ των διαστάσεων που θα έπρεπε, γιατί ειδικά οι Αμερικανοί έχουν συγκεκριμένε θέσει από αυτόν. Αυτή είναι η πιο εύκολη ερώτηση νομίζω που θα μπορούσατε να μου κάνετε σήμερα. Πέρα από την πλάκα τώρα, όταν ε, αναφερθήκαμε στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είπα ότι πρέπει να υπάρχουν στρατιωτικές απαιτήσει ε, μεταξύ του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικού μου του στρατιωτικού επιτελείου, Μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα υπάρχει συμφωνία για τις τεχνικές απαιτήσει, για τις υποδομές αλλά εκεί που δεν φτάσαμε και δεν ε, ασχοληθήκαμε και καθόλου γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι η δική τους αρμοδιότητα ε, ήταν σε τι γεωγραφική κατανομή θα δοθεί για τα κονδύλια. Εμείς είδαμε τις επιχειρησιακές μας προτεραιότητες και είπαμε ότι ο τάδε διάδρομος πηγαίνει στο τάδε σχέδιο εκτακτής ανάγκης, αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα, σας παρακαλώ δώστε τα χρήματα εκεί. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να γίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι δική τους αρμοδιότητα. Τώρα, όσον αφορά την εκτίμηση για το πόσο στοιχίζει. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερι πηγές από τις οποίες θα μπορούσαν να προέρχονται τα χρήματα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επομένως πρέπει να υπάρχει υψηλού επίπεδου πολιτική καθοδήγηση. Αποκλείεται να έρθει από κάτω. Ένα από τις πηγές, μία από τις πηγές που αναφέρεται είναι χώρες οι οποίες εκπαιδεύονται και κάνουν ασκήσεις. Αυτή τη στιγμή πληρώνουν για τις εκπαιδεύσεις και τις ασκήσεις. Και αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τον εξυγχρονισμό των υποδομών. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Μετά, ε, η κάθε χώρα έχει εθνικά σχέδια. Το δεύτερο στοιχείο αυτό. Το τρίτο στοιχείο είναι, αν δείτε, ε, τα πακέτα των ικανοτήτων του ΝΑΤΟ, κάποιος από τους λιμένες, κάποια από τα αεροδρόμια είναι τμήμα του πακέτου κινητικότητας του ΝΑΤΟ και ούτως ή άλλως πρέπει να αναπτυχθεί εντός του ΝΑΤΟ. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ότι ελπίζουμε ότι εν τέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβλέψει κονδύλια στον προπολογισμό για το στόχο αυτό. Από αυτές τις τέσσερις πηγές λοιπόν χρειάζεται πολιτική καθοδήγηση από το υψηλότερο επίπεδο προς τα κάτω γιατί αλλιώς θα δίνουμε μάχη για χρόνια και δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό που είπαμε εμείς ως ένα βήμα που θα μπορούσε να γίνει από πλευράς ΝΑΤΟ, είπαμε ότι θα μπορούσε να γίνει σταδιακά όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, να πούμε ότι θα θέλαμε μέχρι το τέλος του 19 να μπορούμε να έχουμε την ε, Task Force ε, ε, προς την περιοχή επιχειρήσεων του Σαχέλ. Επίσης, μέχρι το 2020 θα ήθελαμε να έχουμε 45.000 ανθρώπους στην ενισχυμένη ε, μονάδα επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Σαχάρας. Επίσης, θα θέλαμε μέχρι το 2028 να μπορούν να μετακινηθούν όλες οι δυνάμεις εντός της Ευρώπης, αλλά αυτή είναι η στρατιωτική σκοπιά. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άμεση σχέση με όλες τις υποδομές αυτή τη στιγμή. Αν όμως καθορίσετε στόχους και δεν τους πετύχετε, τότε θα δείτε πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις συνέπειες. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Διότι ε, τα χρήματα είναι πολλά χρήματα, θα είναι αρκετά δις ευρώ. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι για, για τον Αρκτικό. Ήμουν στην Ισλανδία την προηγούμενη εβδομάδα σε μια επίσκεψη. Στην Αρκτική βεβαίως υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς Κίνας η Κίνα φαίνεται να χρησιμοποιεί κυρίως ε, ήπιες ε, μορφές πίεσης, ενώ ε, οι άλλες πλευρές στρατικοποιούν το, την Αρκτική. Εσείς τι άποψη έχετε για το τι συμβαίνει εκεί, στο βορρά ψηλά. Διότι έχω την εντύπωση ότι κάποιοι σύμμασχοι υποτίμησαν την απειλή την πιθανή απειλή για τις επόμενες δεκαετίες ε, που θα μπορούσε να προέρθει από εκεί. Το ΝΑΤΟ βεβαίως ε, εξετάζει τι συμβαίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εσείς τι άποψη έχετε. Λοιπόν, ένα από τα βήματα τα οποία θα προχωρήσουν στο Υπουργείο Άμυνα αυτήν την εβδομάδα είναι να υπάρχουν διοικητές υπεύθυνοι για τον Ατλαντικό και ταυτόχρονα θα εξετάσουν και την περίπτωση της Αρκτικής. Δεν μπορούμε βεβαίως επισήμως να τα αναφέρουμε αυτά, διότι δεν μπορούμε επισήμως να ασχοληθούμε με την Αρκτική στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η Αρκτική ως ε, μία πλατφόρμα για να παρακολύσει την ενίσχυση και να υπάρχουν εξουσίες. Διότι το ΝΑΤΟ δημιουργείται λόγω ενίσχυσης και την δυνατότητα να έχουμε ενίσχυση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εμεί θεωρούμε ότι η Αρκτική είναι μια πλατφόρμα εξουσίας που θα ε, ε, έχει και παρεμβάσεις στην ε, πολιτική μας και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι κάνει η Ρωσική Ομοσπονδία που στρατικοποιεί την Αρκτική. Για την Κίνα, όπως είπατε, εδώ έχουμε ήπια χρήση δυνάμεων. Η Κίνα πάντα το εξετάζει αυτό από όλες τις προπτικές. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε μακροπρόθεσμα, αλλά προς το παρόν δεν ε, υπάρχει στρατιωτική απειλή για αυτούς. Ε, κυρίως λοιπόν μας ανησυχεί το θέμα ε, της χρήσης ισχύω εδώ. Τώρα, Προηγουμένως αναφέρθηκα σε πρότυπα και τα συζητήσαμε τα πρότυπα. Ένα από τα βασικά πρότυπα του ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιούν ακόμα και οι Ρώσοι, είναι ε, έρευνα και διάσωση στην Αρκτική. Επομένως, είναι αρκετά καλά τα στάνταρ του ΝΑΤΟ. Συνάδελφος από την Πορτοκαλία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε και δύο λόγια για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γερμανία, για αυτά τα σχόλια. Ε, γιατί λοιπόν ε, είναι τόσο σημαντικό αυτό για την Ευρώπη. Απάντηση. Ναι, γιατί οι υπουργοί των κρατών ε, μελών του ΝΑΤΟ θα συμφωνήσουν για τον μηχανισμό ανταπόκρισης πρώτον στον Ατλαντικό και δεύτερον ε, μηχανισμό, κοινό μηχανισμό ε, στήριξης ε, υλικοτεχνικής κτλ. Στην Γερμανία. Στην περίπτωση του Ατλαντικού το κέντρο επιχειρήσεων θα είναι στο Νόρφοξ στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου θα υπάρχει αρμοδιότητα για τις τηλεπικοινωνίες επίσης. Θα υπάρχει βέβαια κάποιος ε, πυρήνας όπου θα διεξάγει τις προετοιμασίες, όμως ε, θα είναι σε λανθάνουσα κατάσταση και μόνο κατόπιν ενεργοποίηση του άρθρου 5 θα ε, κινητοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η προετοιμασία, η εκπαίδευση. Αυτό που δεν θέλουμε όμως είναι να γίνει μόνιμη κατάσταση, διότι όπως σας είπα πρόκειται μόνο για ε, περίπτωση που ενεργοποιηθεί το άρθρο 5. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις? Κυρία Καηλή, εγώ έχω μια ερώτηση, ίσως ε, λίγο πιο πολιτική. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται περιπτώσεις ε, σύγκρουσης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, πιστεύετε πως υπάρχει κάποια ένταση την οποία υποτιμούμε, κάτι που δεν φαίνεται και που θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Ακούσαμε και για τις νέες τεχνολογίες και στο Κοινοβούλιο ασχολούμαστε με αυτές. Θεωρείτε πως ε, υπάρχει απειλή από τα μη επανδρομένα σκάφη ή θεωρείτε πως υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Ναι. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου για αυτό που υποτιμάτε περισσότερο, θα έλεγα πως αυτό είναι οι βρυδικές δραστηριότητες. Οι βρυδικές δραστηριότητες συνδέονται με, ε, με την κυβερνοπηλή και είναι κάτι που υποτιμούμε, πιστεύω. και νομίζω πως υπάρχει ένα ποσοστό αφέλεια στην προσέγγισή μας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πως κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα είμαστε στόχος. όχι απαραίτητα εσκεμένα, αλλά πολλές φορές η από την Κίνα για παράδειγμα, από άλλες χώρες, γίνονται ενέργειες που δεν στοχεύουν απαραίτητα σε εμάς, δεν είναι κάποια εχθρική ε, ενέργεια, όμως ε, υπάρχουν συμβάντα και δεν θέλουμε φυσικά να επαναληφθεί αυτό που έγινε στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν γενικότερα να μην υποτιμάμε τις ε, υβριδικές απειλές. Τώρα, όταν γίνεται λόγος για τεχνητή νοημοσύνη, για αυτόνομα συστήματα τα λοιπά, Εμείς ως ΝΑΤΟ προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στο στρατιωτικό σκέλος αυτής της συνεργασίας και το ερχόμενο έτος θα ε, γίνουν πολλά διότι πιστεύω πως ε, είμαστε ακόμα πίσω. Αν δείτε τι γίνεται με τα μία επανδρομένα σκάφη στο στο Αφγανιστάν θα δείτε πως ε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση, χρειάζεται ενημέρωση και προετοιμασία. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο στην περίπτωση του Αφγανιστάν, αλλά να δούμε και ε, τι θα μπορούσε πιθανά να συμβεί στην Ευρώπη. Και στην περίπτωση της Βαλτικής έχουμε δει αυτά τα ε, σκάφη να μπαίνουν στην επικράτεια των χωρών της Βαλτικής και όχι μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω πως υπάρχουν αρκετά θέματα δεοντολογίας και αρκετά νομικά ζητήματα, οπότε είναι δύσκολο το θέμα. Όμως, όπως ακριβώς με την κυβερνοπηλή και με, τον, ε, ε, με τα θέματα εντοπισμού, νομίζω πως είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, διότι αν δεν ασχοληθούμε εμείς με αυτό, θα χρησιμοποιηθεί από την άλλη πλευρά εναντίον μας. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε με προσοχή τα επιμέρους στοιχεία, με, να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Ξέρω πως είναι δύσκολο το θέμα, όμως ε, χρειάζεται να λυθεί. Θα ήθελα να αντιδράσω πάνω στην ε, ερώτηση που έγινε, ότι τι δηλαδή είναι αυτό που υποτιμούμε. Νομίζω πως ε, καταρχάς υποτιμούμε τους ίδιους τους εαυτούς μας. Υπάρχουν ομάδες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εθνικιστικές, λαϊκιστικές. Και νομίζω πως ως πολιτικοί υποτιμούμε αυτό που μπορεί να γίνει, αυτό που μπορεί να κάνουμε στη συνοχή, είτε στη συνοχή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εντός ΝΑΤΟ, είτε εντός Ηνωμένων Εθνών. Ας δούμε λοιπόν τις ε, ομάδες που έχουν επιθετικές τάσεις ε, προς ε, εμάς και νομίζω πως θα δείτε πως είναι μεγαλύτερες και ισχυρότερες από ό,τι πιστεύαμε. Σας ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση έχω. Μιλήσατε ε, για το ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης εσωτερικών αποφάσεων σε εποχές κρίσης. Τι εννοείτε, πιο συγκεκριμένα θεωρείτε πως ε, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που ενεργούμε. Ναι, αναφέρθηκα νωρίτερα στην ανάγκη ανταπόκρισης. Με αυτό εννοούμε την στρατιωτική ετοιμότητα, τη δυνατότητα να μετακινηθούν δυνάμεις γεωγραφικά και ε, εννοούμε την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Γνωρίζετε πως ε, πολλές φορές χρειάζεται χρόνος μέχρι να ληφθεί μια απόφαση. Θα θέλαμε λοιπόν κάποια στοιχεία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ε, να ανατεθούν ε, στο ΣΑΚΕΡ, για παράδειγμα. Υπάρχει μία task force υψηλού επίπεδου και προς το παρόν το ΣΑΚΕΡ έχει μόνο την δυνατότητα ενημέρωσης και οργάνωσης. Δεν μπορούν δηλαδή να, στή, να ετοιμάσουν ε, μία μονάδα ε, στρατού δεν μπορούν όμως να τη στείλουν πουθενά διότι δεν έχουν την ε, δυνατότητα διοργάνωσης αυτής της μεταφοράς. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών. Και φυσικά θα θέλαμε να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης στρατευμάτων. Όμως στο Συμβούλιο υπάρχουν φωνές που λένε πως το Σάκερ δεν μπορεί να αξιολογήσει την κλιμάκωση μιας ε, κατάστασης και δεν μπορεί επομένως να αναπτύσσει δυνάμεις. Είναι θέμα στρατιωτικής εξουσίας. Μετά, όταν ε, μιλάμε για κινητικότητα, πρέπει να δούμε ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι η κινητικότητα στον αέρα. Αυτό έχει να άμεση σχέση με την ε, κοινή Task Force ανταπόκρισης ε, κρίσεων. Αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ υπάρχει μια ομάδα ανταπόκρισης ε, κρίσεων η οποία σύμφωνα και με αυτά που έχει συζητήσει το Συμβούλιο είναι έτοιμη να αναπτυχθεί και να δραστηριοποιηθεί από τη στιγμή που λαμβάνει την έγκριση από τα κράτη-μέλη. Ορισμένες χώρες έχουν περιθώριο μέχρι και πέντε ημερών για να λάβουν ε, αυτήν την έγκριση, να περάσει από όλα τα διπλωματικά επίπεδα. Και σίγουρα τα κράτη-μέλη έχουν το δικό τους δικαίωμα αποφάσεων, όμως πρέπει να δούμε και πώς συνδέεται αυτή η κοινή ε, task force και πώς λειτουργεί. Η υλικοτεχνική στήριξη λοιπόν, αυτό ακόμα ε, είναι εθνική αρμοδιότητα. Και σε αυτό συγκαταλέγεται και για παράδειγμα το να χρησιμοποιείς πυρομαχικά από ένα άλλο κράτος μέλος. Γι' αυτό σίγουρα θα ε, φέρουμε τους πολιτικούς στα όρια τους, αλλά νομίζω πως πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ, και για την παρουσίασή σας, αλλά και για τις ακριβέστατες απαντήσεις που δώσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς τις απαντήσεις, όπως το κάνατε εσείς σήμερα. Οπότε νομίζω ότι τώρα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον στρατηγό. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Φιλίπ Φλούρι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Παόλο. Οι συνάδελφοι μου ζήτησαν να ολοκληρώσω με τη δικιά μου παρουσίαση τη σημερινή συνάντηση, να κλείσω το θέμα δηλαδή εδώ. Όσοι χάσατε την ανακοίνωση στην αρχή της συνεδρίασης, έλεγε ότι οργανώθηκε ανάμεσα στο κέντρο της Γενέβης για τον δημοκρατικό έλεγχο ε, ενόπλων δυνάμεων και την κοινοβουλευτική συνέλευση. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς όντως τις δύο κοινοβουλευτικές ε, συνελεύσεις ή μάλλον πιο σωστά την κοινοβουλευτική συνέλευση και το κοινοβούλιο να τα βάλουμε μαζί, να γνωριστούν καλύτερα. Αν σκεφτόμασταν πριν από 10 χρόνια θα γινόντουσαν παρόμοιες συναντήσεις για τις απειλές Αφγανιστάν, Ρωσία κλπ. για θέματα ασφάλειας δηλαδή, αλλά τέτοιες συναντήσεις τότε ήταν περισσότερο ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. David και Παόλο. Ήταν ακαδημαϊκού χαρακτήρα λοιπόν. Οι ομιλητές ήταν κυρίως ακαδημαϊκοί. Η αντίληψη που είχαμε για τις απειλές ήταν αυτή στην οποία κατέληγαν τα διάφορα think tanks και όχι οργανισμοί αφοσιωμένοι σε τέτοια ζητήματα και σίγουρα όχι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Φύγαμε λοιπόν από αυτού του είδους τις ε, συναντήσεις γιατί, γιατί μας αποθάρρυναν. Γιατί μία πλευρά κρατούσε το μαστίγιο και άλλη το καρότο. Και δεν καταφέραν οι δύο πλευρές ποτέ να συγκεράσουν τις απόψεις τους. Τώρα από το 2016 και πιο νωρί βέβαια, στην διάρκεια της προετοιμασίας της κοινή ε, δήλωσης, πολλά έγιναν. Και πολλά σωστά έγιναν. Και με ενθαρρύνει πάρα πολύ η σημερινή συνάντηση. Πολλοί από εσά πιστεύω ότι θα νιώσουν ε, πολύ ενθαρρυμένοι και ίσως ακόμα πιο πολύ μετά την αυριανή ημέρα. Όμως δεν λέω ότι γίνονται πάντα τα σωστά πράγματα. Αυτό όμω που λέω είναι ότι ό,τι γίνεται γίνεται με σωστό τρόπο. Δηλαδή, με αυτό εννοώ ότι ακολουθούμε ολόκληρο τον κύκλο για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις απειλές στην ασφαλειά μας. Από τη στιγμή της ενοιολογικής αντίληψης μέχρι την αντίδραση εντοπίζονται απειλές όχι μόνο θεωρητικά, αλλά συζητούμε και για την επιχειρησιακή ικανότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους απειλές. Οπότε, από τη σημερινή συνάντηση, τι κρατάμε. Πρώτα απ' όλα τέτοιες συναντήσεις δεν γίνονται από μόνες τους, οργανώνονται. Άρα είναι προς όφελος όλων των των να οργανώνονται τέτοιου είδους κοινοβουλευτικές, μάλλον διακοινοβουλευτικές καλύτερα ε, διασκέψεις, έτσι ώστε να υπάρξει η καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των απειλών και των δράσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι απειλές. Πάντως από τη σημερινή συνάντηση κρατάω ενθάρρυνση, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει πολλά σωστά και με το σωστό τρόπο. Εγώ προσωπικά Αισθάνομαι ότι τόσα συζητήσαμε σήμερα έχουν πολύ μεγάλη σημασία βέβαια για όλους τους παρόντες. Αλλά πιστεύω ότι αυτές τις ιδέες, τις απόψεις και τα συμπεράσματα θα έπρεπε να τα μοιραστούμε με το ευρύτερο δυνατό κοινό. Γιατί τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει το στάδιο της μεροληψίας εδώ και χρόνια και έχουν φτάσει σε μια κοινή κατανόηση των απειλών, σε μια κοινή κατανόηση του τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις και δυσκολίες τόσο μέσα σε αυτόν τον ευρωατλαντικό χώρο αλλά και εκτός αυτού σε άλλε περιοχές που θα έπρεπε να σταθεροποιηθούν. Συνεπώς, ενθαρρύνω του συναδέρφους της κοινοβουλευτική συνέλευση, να προσπαθούν να βρουν τρόπους να συγκεντρώσουν την σημερινή τεκμηρίωση και να προσπαθήσουν να την δημοσιοποιήσουν. γιατί πιστεύω ότι τέτοιες συζητήσεις μπορούν κάλλιστα να περάσουν στο ευρύ κοινό. Τώρα όσον αφορά εμάς, δηλαδή το κέντρο της Γενέβης για τον δημοκρατικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, εμείς συνεργαζόμαστε και με, την, και με τον ΝΑΤΟ, την κοινοβουλευτική του συνέλευση, δηλαδή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιοι από εσάς αν δεν έχετε ακούσει ξανά για αυτό το κέντρο, να ξέρετε ότι οι χώρες σας εκπροσωπούνται σε αυτό. Μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο www.tcaf.ch Ελβετία λοιπόν, έτσι, πρόκειται για το Διεθνές ε, Κέντρο Δημοκρατικού Ελέγχου Ενόπλων Δυνάμων προωθεί το δημοκρατικό έλεγχο της ασφάλειας, της άμυνας, όπως επίσης και διαχείριση με διαφάνεια αυτών των ζητημάτων. Έχει think tank για τις διάφορες απειλές, για το, τις έννοιες των απειλών αυτών, για παράδειγμα ειρήνη και ασφάλεια ή κυβερνοαπειλές και συνεργάζεται με περιφερειακούς οργανισμούς αλλά και διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε ετοιμάσει διάφορε μελέτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα και συνεργαζόμαστε και με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση πάρα πολύ. Είχαμε ένα σεμινάριο. Συνεπώς, εγώ προσωπικά προσβλέπω και στην δεξιό στο ποτό που θα ακολουθήσει σε λίγο, αλλά και στην αυριανή συνάντηση. Και πραγματικά πολύ χαίρομαι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτό το τομέα. Και παρόλο που δουλεύω σε αυτό το τομέα εδώ και 25 χρόνια, πρέπει να πω ότι δεν ήμουνα τόσο καλά ενημερωμένος όπως είμαι τώρα. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ιδέες και τις σκέψεις σας και προσβλέπω στη συνέχεια αύριο. Κύριε Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από την Ελβετία και το κέντρο της Γενέβης για το Δημοκρατικό Έλεγχο Ενόπλων Δυνάμεων είναι ότι διατηρείται την ισορροπία μεταξύ των διεθνών δυνάμεων. Οπότε, όντω και θέλετε κάτι να ρωτήσετε, γιατί έκλεινα τώρα. Εντάξει, παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα σχόλιο έχω να κάνω και μια παρατήρηση. Σαφώς το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συνεργαστούν πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Μπορεί να είναι περίπλοκο, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση πάνω απ' όλα. Απαιτεί όμως και μη ευρωπαϊκές χώρες στο ΝΑΤΟ να πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν έρχομαι στο θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία θα υπάρξει εφόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ υπάρχει. Υπάρχει διάλογος ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς ε, πολιτικούς. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε τι επίπεδο γίνεται ο διάλογος αυτός ανάμεσα στους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Αμερικανούς. Γιατί για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να πείσουμε τους Αμερικανούς και τους Αμερικανούς πολιτικούς ότι δεν είναι σημαντικό μόνο το ΝΑΤΟ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τους. Πρόεδρος, και εγώ θα έλεγα ότι ναι, συνεχίζεται ο διάλογος, δεν έχει σταματήσει και είναι νομίζω πολύ καλό αυτό που λέτε. Εγώ δεν ξέρω αν πιστεύουν ή όχι οι Αμερικανοί στην Ευρώπη. Αυτό όμω που μπορώ να πω είναι ότι χρειαζόμαστε ένα τον άλλον, ότι είμαστε σύμμαχοι, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Ο διάλογο αυτό, οι ερωτήσεις και απαντήσεις που είχαμε σήμερα παρόλο που κάλυψαν λίγο πολύ όλες τις πτυχές που μας απασχολούν, αποτελούν περισσότερο τροφή για σκέψη, αλλά και τροφή για κατάρτιση πολιτικής και για δράση, όταν διαπιστώνουμε ότι κάπου έχουμε μείνει πίσω. Πρέπει να βρούμε νέες λύσεις. Είναι έτσι κι αλλιώς κάτι το οποίο συνεχώς συνεχίζεται στην πολιτική, δεν τελειώνει ποτέ. Σας ευχαριστώ πάντως και σας ευχαριστώ όλους για την προσέλευσή σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρουσία σας εδώ δείχνει και το γεγονός ότι οργανώθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει πόσο μεγάλη σημασία δίνει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στη διπλωματία σε αυτά τα θέματα. Αν λοιπόν υπάρχουν ζητήματα οι πολιτικοί που φροντίζουν να ακουστεί η φωνή των πολιτών θα αναλάβουν δράση. Η σημερινή λοιπόν συζήτηση ήταν υψηλού επίπεδου πραγματικά. Η κυρία Κέτε Μίλλερ είπε πριν φύγει από δύσκολες ερωτήσεις. Δύσκολες ερωτήσεις που απαντήθηκαν Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για παρετέρω βελτίωση των σχέσεών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Άλλη είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουμε εδώ. Καλή αρχή. Οπότε αγαπητέ Πρόεδρε, αύριο θα επισκεφθούμε τη στρατιωτική ικανότητα σχεδιασμού. Στις 9 θα συναντηθούμε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Renaissance και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και στην δεξίωση στο Ισόγειο, στο Σαλόνι 6. Είναι δεξίωση που προσφέρει ο Αντιπρόεδρος Πάσκου εκ μέρους του Πρόεδρου Ταγιάννη. Σας προσκαλούμε λοιπόν εκεί. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίστε να φροντίσετε για την ισορροπία όπως κάνουν οι Ελβετοί έτσι καλώς. Ευχαριστώ πολύ.